Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών και παρακαλώ να καθίσετε όλοι. Όσοι είστε πίσω-πίσω, παρακαλώ, καθίστε. Να ξεκινήσουμε αυτή τη σημαντική συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών. Καταρχήν, Θα ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου Λαμασούρ και των ε, άλλων ε, παλαιότερων αντιπροέδρων που δεν μπορούσαν να είναι σήμερα παρόντες και άρα πρέπει εγώ να προεδρεύσω. Παρακαλώ όλους να καθίσετε. Η συζήτηση όσον αφορά τις εκτιμήσεις ε, μπορεί να γίνει και εκτός της αιθούσης. Συνάδελφοι, έχουμε πάρα πολύ σημαντική συζήτηση σήμερα το πρωί. Η Σιδόνια θα μας οδηγήσει σε αυτή τη συζήτηση. Ας ε, δούμε πρώτα για το σημείο 1. Υπάρχουν θέματα για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Ανακοινώσεις Προέδρου ούτε. Μόνο να σημειώσουμε τις αποφάσεις ε, στο 10 Μαρτίου των συντονιστών. Σημείο 4, που είναι το κύριο σημείο υποσυζήτηση σήμερα, είναι η δημόσια κρόση για την χρηματοδότηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Όπως γνωρίζετε, η ανατολική εταιρική σχέση ξεκίνησε το 2009. Είναι μια πρωτοβουλία πολιτικής που συμπληρώνει την εξωτερική πολιτική της Ένωσης προς την Ανατολική Ευρώπη και τον Νότιο Κάυκασο, ε, χώρες ε, που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γετνίασης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει περίπου 2,8 δις ευρώ ώστε να προωθήσει τι απαραίτητε συνθήκες για να επιταχυνθεί η πολιτική και η οικονομική ολοκλήρωση ανάμεσα στην, ε, ανάμεσα στην Ένωση και διάφορες ε, χώρες ε, όπως η Μολδαβία, η Ουκρανία η, και, και άλλες χώρες της περιοχής. Εμείς σήμερα κάνουμε μια ανακρόαση για τη χρηματοδότηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης και η ιδέα είναι να έχουμε μια γενική εικόνα για αυτό το περίπλοκο ζήτημα, την εφαρμογή των, την υλοποίηση και την εφαρμογή την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων και αυτοί που εφαρμόζουν τα προγράμματα θα είναι εδώ για να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα επιτόπου. Εξ ονόματο τη Επιτροπή Προπολογισμού, θέλω να καλωσορίσω του εκπροσώπου τη Κομισιόν, του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θα μα εξηγήσουν πώ λειτουργεί η χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή ε, ανατολικής εταιρική σχέσης και έχουμε και εκπροσώπους διαφόρων ε, ομάδων ε, προβληματισμού που θα μας πούν τη γνώμη τους για αυτή την σημαντική πολιτική πρωτοβουλία. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στη Σιδωνία ως εισηγήτρια για να μας παρουσιάσει πιο λεπτομερώς πώς θα προχωρήσει η σημερινή ακρόαση. Σιδωνία. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην σημερινή πρωινή συνεδρία της Επιτροπής Προπολογισμών που ε, θα εστιάσει στο θέμα της χρηματοδότησης της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Σαφώς όταν δει κανείς τον ορισμό, τα πράγματα φαίνονται απλά. Η ε, ανατολική εταιρική σχέση είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς έξι ανατολικούς εταίρους Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία. Και ο στόχος είναι να βελτιωθούν οι διμερείς αλλά και οι πολυμερείς σχέσεις ανάμεσα στις χώρες αυτές και την Ένωση. Η ιδέα είναι να δεσμευθούν ε, οι εταίροι στις αρχές ε, του διεθνούς δικαίου και των διεθνών αξιών συμπεριλαμβανομένων ε, το κράτος δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και η πρόθεση της βιώσιμης και ορθής διακυβέρνησης. Η εταιρική σχέση δεν είναι βέβαια αυτός σκοπός. Θέλει να παρέχει τα θεμέλια για νέες συμφωνίες ε, σύνδεσης ανάμεσα στην Ένωση και τους εταίρους εκείνους που έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο προς τις αρχές και τις αξίες αυτές που αναφέραμε. Θα εστιάσουμε την προσοχή σήμερα στο θέμα της ε, χρηματοδότησης αυτής της πρωτοβουλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, κρατήσει 2,8 δις για την εταιρική σχέση αυτή για την περίοδο 2009 με 2013. Και πρέπει να πούμε ότι τώρα βρισκόμαστε ακόμη σε διαπραγματεύσεις, ακόμα διαπραγματευόμαστε μάλλον το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οπότε δεν γνωρίζουμε τι χρήματα θα έχουμε στη διάθεσή μας ε, στο μέλλον. Ωστόσο έχουμε κάποιες ιδέες υπό τη μορφή της αρχικής πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των γενικών κατευθύνσεων ε, της διάσκεψης κορυφής του Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να εξηγήσω τα κίνητρα, τα αίτια που μου οδήγησαν εμένα στο να συγκαλέσουμε αυτή τη σημερινή συνεδρίαση. Είναι, πρόκειται για μια προσωπική μου εμπειρία. Πέρυσι προσεκλήθην από το Ινστιτούτο Ρομπέρ Σουμάν σε μια διάσκεψη, σε μια εκδήλωση, μια συνάντηση με νέους ε, ηγέτες της ε, αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο προωθεί το Ινστιτούτο Ρομπέρ Σουμάν, ε, λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια μέσα στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ονομάζεται «Ηγεσία προς τη Δημοκρατία». Η ιδέα είναι να προετοιμαστούν νέοι υποψήφοι για μελλοντική και πολιτική σταδιοδρομία και εν τέλει έτσι ώστε να βοηθηθεί η δημοκρατική μετάβαση στη Λευκορωσία. Μου ζητήθηκε να ενημερώσω τους συμμετέχοντες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προς τη Λευκορωσία, αλλά γενικότερα προς τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Προετοιμαζόμενοι γι' αυτό, για αυτή την εκδήλωση, διαπίστωσα ότι η χρηματοδότηση είναι πολύ διασκορπισμένη και η ενημέρωση σχετικά με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση εξαιρετικά περίπλοκη. Είναι περίπλοκη γιατί η ανατολική εταιρική σχέση στην ουσία είναι μια ομπρέλα που συνδυάζει διάφορα προγράμματα και δημοσιονομικά μέσα που αφορούν όχι μόνο αυτές τις έξι χώρες, αλλά και πολλές άλλες χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να εκτιμήσουμε λοιπόν τα ποσά που χορηγούνται σε κάθε μια από αυτές τις χώρες ε, είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και ακόμα πιο δύσκολο είναι να αξιολογήσουμε την χρήση αυτών των χρημάτων επιτόπου. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι θα πρέπει εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμού να έχουμε μια καλά διαρθρωμένη συζήτηση για τα χρήματα που στόχο έχουν να χρηματοδοτήσουν την ανατολική εταιρική σχέση τώρα και με την προοπτική του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου τι μπορούμε να μάθουμε καλύτερα και τι μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε καλύτερα στο επόμενο πολιετές. Θέλουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Εγώ φυσικά εστιάζω στα ερωτήματα που θεωρώ πως συνδέονται με τη δουλειά της Επιτροπής Προπολογισμού. Καταρχήν ένα πολύ βασικό, πόσα χρήματα ε, ε, πηγαίνουν στις χώρες της ε, εταιρική σχέσης, ποια μέσα είναι αφιερωμένα στους έξι συμμετέχοντες και τέλος ποια είναι η χρήση αυτών των χρημάτων και εκμεταλλευόμενοι τους διάφορους συμμετέχοντες σε αυτή την εκδήλωση να μάθουμε από τις εμπειρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ΜΚΟ και άλλων οργανισμών όταν εφαρμόζουν τη βοήθεια χρησιμοποιούν τη βοήθεια που ε, κατευθύνεται στις χώρες αυτές και πώς ε, οι συμμετέχοντες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα διδάγματα που αποκομίσαμε για τη χρήση των χρημάτων τα επόμενα 7 χρόνια. Ας εστιάσουμε την προσοχή στο πρόγραμμα για το σημερινή συνεδρίαση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με όσους ε, χρησιμοποιούν τα χρήματα επιτόπου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το κομμάτι το κάνει η Γενική Διεύθυνση και με χαρά βλέπω εδώ τον κύριο Μάρκος Κορνάρο που είναι ο αναπληρωτής διευθυντή, γενικός διευθυντής της διεύθυνσης και ε, καλύπτει και την Ευρω... Ε, γυτνίαση e <clears throat> των... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό και ευπρόσδεκτο ότι ο κύριος Χάιντς Χόλμπερτ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι επικεφαλής είναι αρμόδιος. Α, δεν είναι εδώ. Α, είστε πολύ ταπεινοί, είστε τόσο μακριά. Ε, είμαι χαρούμενη που είναι εδώ σήμερα ο κύριος Χάρη Όλμπερ, εκπροσωπώντα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να μα πει περισσότερα για το τι μέσα χρησιμοποιεί στη συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Ιτρικής σχέση και όταν θα έχουν γίνει αυτέ οι παρουσιάσει. Θα έχουμε και μια κριτική άποψη από δύο ακαδημαϊκούς που εργάζονται για το θέμα ε, και συγκεκριμένα από τον κύριο Όλα που είναι διευθυντής ανατολικών σπουδών ε, στην Πολωνία και θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσε να μας μιλήσει κάπως περισσότερο για αυτή την αρχή more for more, περισσότερα για περισσότερα για το εμάς του προπολογισμού είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς πληρώνεις περισσότερα για περισσότερη δημοκρατία, πώς μετράτε αυτό, πώς ποσοτικοποιείται και η άλλη ε, παρουσίαση θα γίνει από την κυρία Γιολάντα Τασνίνκα που είναι από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, του Πανεπιστημίου του Λούτς και θα μοιραστεί μαζί μας ε, τη δική της εντύπωση για την εφαρμογή του προγράμματος επιτόπου και πιο συγκεκριμένα στην Ουκρανία. Με χαρά επίσης θα ακούσουμε και την προοπτική μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης γι' αυτό θα μας μιλήσει η κυρία Άννα Κριστίνα Λίνκα, διότι όταν προετοιμαζόμουν για αυτή τη συζήτηση ανακάλυψα ότι το Conrad Αντενάουερ Stiftung είναι ένα σημαντικός δικαιούχος αυτών των ε, ε, κονδυλίων το Ίδρυμα Conrad Αντενάουερ ε, και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι σημαντική αυτή η συμβολή. Τέλος, ο κύριος ε, Τίμπελ θα μας, δώσει μια, θα μας ε, μιλήσει για το μέλλον, που είναι επικεφαλής ε, του τμήματος της Ανατολικής εταιρική Σχέσης στην Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία. Α, είστε πολύ πίσω, δεν σας είχα δει. Ελπίζω πως θα είναι αισιόδοξο το θα μας πείτε για το μέλλον. Θα ήθελα επίσης ε, να καλωσορίσω και όλους όσους δεν απαριθμούνται εδώ που είναι στο ακροατήριο και αντιπροσωπεύουν ε, διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την ε, ανατολική ιατρική σχέση και έχουμε επίσης χρόνο, ελπίζω, ελπίζω πως θα έχουμε αρκετό χρόνο, να ακούσουμε και να συζητήσουμε και με το ακρατήριο. Αν μου επιτρέπετε να προτείνω να γίνει μια συζήτηση στο τέλος, ώστε να συζητήσουμε όλα τα θέματα Ελπίζω πως θα είναι πολύ ζωντανή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Uh, Ωραία. Οπότε παρακαλώ τον πρώτο ομιλητή να ξεκινήσει. Είναι ο κύριος Μάρκος Κορνάρο. Δεν ξέρω αν έχουμε λίστα προβλήματα με τις προβολές. γιατί αλλιώ φοβόμουν πως θα έπρεπε να κοιτάζουμε το τυπωμένο έγγραφο, αλλά φαίνεται ότι όλα είναι εντάξει. Χαίρομαι που υπάρχει αυτό, αυτή η δυνατότητα να σας δείξω. Νομίζω πως είναι καλύτερα να έχετε και τα και τα slides φαίνεται πώς κάνουμε ορισμένα πράγματα που και μετά θα μιλήσω για ορισμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ελπίζω η παρουσίαση να επιβεβαιώσει ότι για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες όλων των ε, τμηματικών και κάπως κατακαιρματισμένων ε, προσπαθειών και μέσων μας. Βεβαίως ε, βλέπετε ότι οι χώρες που είναι με πράσινο δεξιά των χωρών της Ένωσης και, της Ένωσης και, των, και των χωρών που είναι υποψήφιες είναι οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Είναι λοιπόν αυτές οι έξι χώρες. Μπελαρούς, Μολδόβα, Ουκρανία, Ουκρανία είναι πολύ κοντά ε, στην Ευρώπη και μετά οι τρεις χώρες του Καυκάσου που είναι λίγο μακρύτερα. Αλλά δεδομένου και του ε, ενδεχόμενου ρόλου της Τουρκίας ε, για τα μελλοντικά καθήκοντα της Ένωσης, άρα και αυτές οι τρεις χώρες είναι κοντά μας. Εδώ βλέπετε τώρα τον Επίτροπο Φίλε που είναι αρμόδιος για τη λειτουργία των διαφόρων μέσων. Μια επισκόπηση λοιπόν της ανατολικής εταιρικής σχέσης και των μέσων της. Οι επόμενες διαφάνειες θα εξηγήσουν τι σημαίνει το μέσο αυτό και πώς λειτουργεί το μέσο, το ευρωπαϊκό μέσο για την ανατολική γειτονία και τα άλλα μέσα που συνθέτουν την εικόνα. Εδώ βλέπετε πόσο κατακερματισμένες είναι οι προσπάθειές μας. Οι δύο κόκκινες στήλες είναι κυρίως ε, γεωγραφικώς λειτουργούντα όργανα, ενώ οι άλλες στήλε είναι κλαδικές πρωτοβουλίες ή θεματικές. Τις χρησιμοποιούμε στο μέτρο του δυνατού για να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται τη βοήθεια που δίνουμε σε αυτές τις χώρες. Πρώτα απ' όλα, τι είναι το μέσο για την ευρωπαϊκή γειτονία και εταιρική σχέση, τι κάνει λοιπόν, προσπαθεί να βοηθήσει τις χώρες αυτές είναι σε φάση αναθεώρησης και θα αποκληθεί στο μέλλον ανατολικό μέσο εταιρικής σχέσης. Είναι 2,8 δις για την προηγούμενη περίοδο προοπτικών. Σημειώνω ότι το ποσό αυτό περιέχει και δύο συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις που αποφασίστηκαν από την Ένωση, συνολικά 500 εκατομμυρίων. Τι χρηματοδοτούμε με το μέσο αυτό. Τα δύο τρίτα δίδονται διμερός μέσω συμφωνιών που συνάπτουμε με τις χώρες αυτές και που μεταφράζονται σε αιτήσια πρόγραμμα δράση. Έχουμε όμως και ένα περιφερειακό πρόγραμμα. Πολλά από όσα γίνονται στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης περιέχονται σε αυτό το πρόγραμμα. Δια περιφερειακή συνεργασία. Έχει ένα μεγάλο μέσο που καλύπτει και τον Νότο και την Ανατολή το κυριότερο είναι το μέσο για την ε, γειτονιακή για τις γειτονιακές επενδύσεις όπου βοηθάει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και το Erasmus Mundus με το, με το οποίο χρηματοδοτούμε επιπλέον κινητικότητα των φοιτητών και η διαμεθοριακή συνεργασία μας βοηθάει να χρηματοδοτήσουμε ενέργειες μεταξύ χωρών κρατών ε, μελών που έχουν κοινά σύνορα με χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και τις όμορες αυτές χώρες. Πώς εφαρμόζονται. Ένα τμήμα περνάει μέσω στήριξη των προϋπολογισμών των ε, χωρών που αποφελούνται και ε, ορισμένες άλλες χρηματοδοτήσεις γίνονται μέσω συμβολέων με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, με διμερεί συμβόλαια, με συμφωνίες συμβολής για κάποια προγράμματα και μέσω διεθνών οργανισμών. Και για τα λοιπά είναι ο συνδυασμός επιδοτήσεων με δάνεια από τους δανειοδοτικούς οργανισμούς της Ένωσης. Ποιοι επωφελούνται από αυτά τα τρία περίπου σε μεγάλο βαθμό δημόσιοι οργανισμοί αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιωτικοί φορείς, όπως ε, θα πω και η κοινωνία των πολιτών στις έξι αυτές χώρες. Δεν θα μιλήσω για τη δημοσιονομική στήριξη. Ίσως προκύψει στη συζήτηση κατόπιν. Οποτεδήποτε συζητάμε τον προϋπολογισμό των δημοσίων οργανισμών ή της δημόσιας διοίκησης, προσπαθούμε να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους για περαιτέρω προσέγγιση της νομοθεσίας τους, των διαδικασιών τους, στα αντίστοιχα του κοινοτικού κεκτημένου. Και εφόσον διαπιστώσουμε ότι έχουν γίνει οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, παρέχουμε αυτή τη στήριξη στήριξη στην κοινωνία των πολιτών. Ήταν ε, τμήμα της πολιτικής ανατολικής γειτονίας εξ αρχής, αλλά ενισχύθηκε στα πλαίσια των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών, διότι καταλάβαμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε όχι μόνο τις κυβερνήσεις, περισσότερο τις κυβερνήσεις, αλλά να έχουμε εταιρική σχέση και με τους λαούς κύριος φορέας γι' αυτό, για μια δική μας οργάνωση, είναι να διασφαλίσουμε ότι ευρύτερα η κοινωνία των πολιτών, ομάδες πολιτών, εποφελούνται. Βοηθάμε διάφορες πρωτοβουλίες που να μας επιτρέπουν και να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι γίνεται, αλλά και να την χάνουν οι πρωτοβουλίες μας περισσότερη στήριξη από την κοινή γνώμη για να αποκτήσουν περισσότερες δυνατότητες αποτελεσματικότητας. Έχουμε λοιπόν το μέσο για την κοινωνία των πολιτών που είναι τμήμα της πιο διαρθρωμένης προσέγγισης για τις ανταλλαγές φοιτητών, για παράδειγμα, και όπως λέει εδώ το τελευταίο σημείο, το συμπληρώσαμε χάρη και στην ισχυρή πρωτο... Ε, ενίσχυση στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτό το ευρωπαϊκό μέσο για την ε, δημοκρατία που μας βοηθάει ε, να στηρίξουμε και μη κυβερνητικές οργανώσεις και τη δημιουργία κομμάτων. Λοιπόν, αναφέρθηκε ήδη στην εισαγωγή η έννοια του περισσότερα για περισσότερα. Υποθέτω ότι θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Για μας τι σημαίνει αυτό στα πλαίσια του αναθεωρημένου μέσου για την πολιτική γειτονία. Πιστεύουμε ότι οι χώρες αυτές που κάνουν μια ειλικρινή και ουσιώδη προσπάθεια για εμβάθυνση της δημοκρατικής μετάβασης, ε, της συνταγματικής αλλαγής, ε, θα πρέπει να έχουν ε, μία περαιτέρω ενθάρρυνση, δηλαδή συμπληρωματική χρηματοδότηση για να ενισχύσουν είτε το κόστος των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και κάποιες προσπάθειες εμβάθυνσης οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα συνολικό που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης να ενισχύει όπου έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτές τις χώρες. Είναι λοιπόν ένα συμπληρωματικό κίνητρο. Στον πρώτο γύρο αυτής της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης βοηθήσαμε έτσι περισσότερο τη Μολδόβα, την Γεωργία και την Αρμενία ενώ για τις άλλες τρεις χώρες Ουκρανία και βέβαια Μπελαρούς εδώ δεν δόθηκαν χρηματοδοτήσεις, αλλά και το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο έχει πιστοδρομήσει από ορισμένες πλευρές της δημοκρατικής μετάβασης. Έτσι λοιπόν επιβραβεύουμε τη σχετική πρόοδο σε κάποιες χώρες. Πιο συγκεκριμένα τι κάναμε στα πλαίσια του προγράμματος περιφερειακής συνεργασίας ε, άμεσα ενισχύοντας την ανατολική εταιρική σχέση. Είχαμε πέντε εμβληματικά προγράμματα για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να συνεργαστούν μεταξύ τους και να αναπτύξουν θετικές πρακτικές σε διάφορους τομείς. Η πρώτη εμβληματική πρωτοβουλία Η πρώτη λοιπόν είναι ε, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης συνόρων για να ενισχύσουμε την ε, ασφάλεια, να μειωθεί το λαθρεμπόριο και η εμπορία προσώπων. Εδώ δώσαμε 44 εκατομμύρια. Δεύτερη πρωτοβουλία εμβληματική το μέσο για τις ε, ΜΜΕ για να βοηθήσουμε σε μεγάλο βαθμό τον ιδιωτικό τομέα και συμβουλές της επιχειρήσεις και αύξηση της επιχειρηματικότητας, ε, δάνεια προς τράπεζες, όπου συμμετέχουν οι επιχειρηματικές κοινότητες από τις δύο πλευρές τρίτη εμβληματική πρωτοβουλία Innogate είναι τα αρχικά στα αγγλικά για την ενοποίηση των αγορών ηλεκτρισμού, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, αύξηση της ε, χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πολύ καλό παράδειγμα επέκτασης των δικών μας πολιτικών για την ενοποίηση των αγορών ενέργειας και ηλεκτρισμού Επέκταση λοιπόν, όχι μόνο διμερός, αλλά και πολυμερός, περιφερειακά, σε αυτές τις χώρες, ούτως ώστε να γίνει μια βιώσιμη πραγματικότητα. Τέταρτη εμβληματική πρωτοβουλία για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ αυτών των χωρών και της Ένωσης για την πρόληψη, την ετοιμότητα και ανταπόκριση σε θεομηνίες. Και πέμπτο, όλες οι χώρες αυτές συμμετέχουν σε μια προσπάθεια για καλύτερη περιβαλλοντική διακυβέρνηση, ε, κλιματική αλλαγή, δασονομία και γενικότερα ε, σε επίπεδο δήμων περιβαλλοντική διαχείριση. Όπως ε, είπα και νωρίτερα, αξιοποιήσαμε το μέσο επενδύσεων της πολιτικής γειτονίας στις χώρες αυτές της ανατολικής γειτονίας με πολύ εντυπωσιακό πρώτο, περίπου 700 εκατομμύρια συνεργαζόμενοι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την ανα, ε, και ανάπτυξη και άλλους ε, δανειοδοτικούς οργανισμούς σε διάφορους τομείς. Τι κάνει λοιπόν αυτή, αυτό το μέσο επενδύσεων βοηθάει τη χορήγηση δανείων, επιδοτώντας ένα τμήμα τους. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να πω και σε εσά που είστε τμήμα της αρχής επί του προπολογισμού. Αυτός ο συνδυασμό έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Ένα ευρώ από επιδότηση από τον προπολογισμό της Ένωσης προκαλεί 30 ευρώ συμπληρωματικής επένδυσης και θα σας πω ε, πιο συγκεκριμένα πώς λειτουργήσε αυτή η προσπάθεια στις σχέσεις με την Τράπεζα Επενδύσεων. Διαμεθοριακή συνεργασία. Περαιτέρω συγκεκριμένη δράση για αυτήν την ε, ανατολική σχέση. Στόχος μας να υπάρχει μια ενιαία χρηματοδότηση ούτως ώστε οι περιθωριακές περιοχές της Ένωσης στη Φιλανδία, την Πολωνία και άλλες ανατολικές χώρες της Ένωσης να μπορούν να συνεργαστούν διαμεθοριακά με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γεωργία και τις χώρες του Καυκάσου, τις άλλες χώρες του Καυκάσου. Μέσω ενός ε, μεγάλων διαστάσεων προγράμματος που επιδιώκει οικονομικές και κοινωνικές ανταλλαγές βοηθάμε τη συνεργασία από άτομα σε άτομα, από άτομο σε άτομο. Θέλουμε η διάβαση των συνόρων να είναι πιο ασφαλής αλλά και πιο άνετη. Πώς ε, έχει τώρα η δημοσιονομική δομή αυτού του προγράμματος. Τα μισά είναι μέσω της γειτονίας αυτής και τα άλλα μισά είναι συμβολές από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο. Εδώ βλέπετε τις προσπάθειες που κάνουμε να βοηθήσουμε τους ανατολικούς εταίρους μέσω άλλων πρωτοβουλειών που λέγονται η διδημοποίηση, το ΤΑΕΞ και το ΣΥΓΜΑ. Τι σημαίνει η διδημοποίηση. Οι δημόσιοι οργανισμοί των κρατών μελών συνεργάζονται με δημόσιους οργανισμούς από τις ε, χώρες αυτές. TAEX ε, σημαίνει πιο βραχυπρόθεσμη χορήγηση ε, τεχνογνωσίας. Οι χώρες μέλη δηλαδή προσπαθούν να βοηθήσουν αυτές τις χώρες, πώς να βοηθήσουν το δασμολογικό τους καθεστώς, ε, φυτο-υγειονομικές ε, βελτιώσεις και ιδιαίτερα οι διοικήσει των ε, νεωτέρων κρατών μελών, των πιο πρόσφατων κρατών μελών που πρόσφατα προσαρμόστηκαν στο κοινοτικό κεκτημένο, βοηθούν τις χώρες από αυτή την περιοχή για να πράξουν κάτι παραπλήσιο. Και σίγμα είναι κάτι ε, ανάλογο με αυτό που κάνουμε με τον ΟΣΑ, δηλαδή βέλτιθες πρακτικές για τη διοίκηση, τη δημόσια διοίκηση και την ε, διαχείριση της οικονομίας γενικότερα. Καταλήγοντας, Ποια άλλα μέσα έχουμε για τις χώρες αυτές. Έχουμε διάφορες κλαδικές δυνατότητες από την αναπτυξιακή συνεργασία, από το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας, προστασία περιβάλλοντος, επενδύουμε στο λαό, επισητιστική ασφάλεια και ε, ένα τμήμα για τη μετανάστευση. Πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε αυτά που χορηγούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε και τοπικά προγράμματα ενίσχυσης δραστηριοτήτων εκδημοκρατισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όπου είναι πολύ δύσκολο αυτό όπως το Μπελαρούς, λαμβάνουν κεντρικές χρηματοδοτήσεις το μέσο για την ε, σταθερότητα που ε, το διαχειρίζεται η υπηρεσία εξωτερικής δράσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει μερικές παγωμένες διενέξεις που δυστυχώς παραμένουν όπως την ορεινή Καραμπαχία ή την ε, υπερδνηστερία. Και έχουμε ουσιώδη προσπάθεια για την πυρηνική για την συνεργασία πυρηνικής ασφάλειας. Προωθούμε λοιπόν και την πυρηνική ασφάλεια και βοηθάμε την ολοκλήρωση του καθαρισμού του Τσιαρνόμπλου. Οπότε, νομίζω σας ενημέρωσα για τις κυριότερες προκλήσεις που διαπιστώσαμε στην προσπάθεια εφαρμογής αυτής της πλειάδας μέσων και όλα αυτά τα έχουμε συμπεριλάβει στις προτάσεις που κάνουμε για την αναθεώρηση του μέσου για την ευρωπαϊκή σχέση γειτονία. Για το ευρωπαϊκό μέσο γειτονία. Αυτή μας η πολιτική μας επιτρέπει να ε, συντονίσουμε καλύτερα την πολιτική με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Αλλά βέβαια πολλά παραμένουν ανοιχτά. Με κάθε χώρα εξετάζουμε πολύ προσεκτικά πόσο μπορεί να συμβάλλει η Ένωση για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθειά μας συνδέεται άμεσα με τους στόχους μας. Βεβαίως ε, ομολογώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα για να συμμετέχουν περισσότερο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Βεβαίως ε, η κοινωνία των πολιτών είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να ενισχύσουμε την εταιρική σχέση με τους λαούς. Και εδώ θα μπορούσαμε ακόμη να βελτιώσουμε. Περαιτέρω τις δραστηριότητές μας. Κατά την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο έχει αλλάξει πολύ ο ρόλος της Ρωσίας και θα δείτε ότι η αναθεωρημένη πρότασή μας αντανακλά την πεποίθησή μας ότι θα πρέπει να ε, εμπλακούμε πολύ περισσότερο με τη Ρωσία ως ε, συνεργάτη μας, αλλά όχι στρατηγικού εταίρου. Είναι ενδιαφέρουσα η εμπειρία και ορισμένα διμερή προγράμματα με τη Ρωσία διακόπησαν κατά αυτή την περίοδο διότι ε, τους ενδιαφέρει περισσότερο η περιφερειακή διάσταση της συνεργασίας. Η προσπάθεια αναθεώρησης ε, είναι στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας ε, απλοποίησης και εναρμόνισης ε, των πολιτικών μας και του προγραμματισμού χορήγησης της βοήθειάς μας. Όπως είπα, έχουμε εισαγάγει ισχυρότερη διαφοροποίηση και την προσπάθεια του περισσότερα για περισσότερα, αλλά και αυτό πρέπει να εκλεπτυνθεί και να προσαρμοστεί περισσότερο όσο συλλέγουμε πείρα και όσο διαπιστώνουμε πώς απορροφούν οι χώρες αυτές τις ε, χρηματοδοτήσεις μας. Η δυνατότητα γενικότερα απορρόφησης είναι καλή. Με ικανοποίηση να σας ενημερώσω ότι μέχρι στιγμής δεσμεύσαμε το 100% της χρηματοδότησης και εκταμιεύσαμε πάνω από 99% την τελευταία επταετία, αλλά αν το εξετάσουμε πιο λεπτομερώς, θα διαπιστώσουμε ότι για κάποια προγράμματα, σε κάποιες χώρες, υπήρξαν κάποια προβλήματα απορρόφησης και γι' αυτό θέλουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μας, ελπίζοντας να τα πάμε ακόμη καλύτερα στα επόμενα χρόνια. Και για την δημοσιονομική στήριξη ε, το 50% περίπου της ενίσχυσης εδώ έχει περάσει στους ε, κρατικούς προϋπολογισμούς. Ενισχύουμε επίσης τις ε, απαιτήσεις μας για προϋποθέσεις καλύτερης διαφάνειας, καλύτερης εφαρμογής του προϋπολογισμού εμπλέκοντας την κοινωνία των πολιτών και καταλαβαίνοντας καλύτερα τα μητρώα πολιτικής που σχετίζονται με τα προγράμματα αυτά. Νομίζω ότι και εδώ τα πάμε αρκετά καλά, αλλά και αυτός είναι ένας τομέας που δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. Όπου δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. Τέλος, καλύτερες, ε, καλύτερη προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των διαφόρων ε, χρηματοδοτικών μέσων εξακολουθεί να είναι πρόκληση. Η απάντηση θα προκύψει μέσω καλύτερης συνεργασίας ε, δικής μας με την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης και καλύτερη συνεργασία με τις επιτόπου αντιπροσωπείες μας που είναι σε θέση να εξετάσουν την πλήρη γκάμα των δραστηριοτήτων αλλά και περισσότερες προσπάθειες επεξήγησης του πώς λειτουργούν τα μέσα στους εταίρους μας όλους τους εμπλεκομένους φορείς τις χώρες αυτές. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε κάποιες από αυτές τις προκλήσεις. Καλό θα ήταν η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας να εφαρμόσει το θεματολόγιο για την αλλαγή που προτείναμε πέρυσι και που ενεκρίθη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όπου θέλουμε να είμαστε πιο στόχο προσιλωμένοι για να επιτύχουμε τη μέγιστη επίπτωση και τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ελπίζω λοιπόν κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, ήδη από το 2013, να έχουμε λιγότερες τομεακές παρεμβάσεις με περισσότερα αποτελέσματα. Είχαμε μια ευρία αναθεώρηση το 2011 του μέσου αυτού, όπου εισαγάγαμε την αρχή της διαφοροποίησης και του περισσότερο για περισσότερα. Ήδη επίσης στην αναθεώρηση αυτή αντιληφθήκαμε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε περισσότερο την κοινωνία των πολιτών και νομίζω ότι και εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε τους καρπούς της νέας μας προσπάθειας. Επίσης αυξήσαμε τα καινοτόμα μέσα μέσω αυτού του συνδυασμού χρηματοδοτήσεων με την Επιτροπή Εξωτερικών, ε, Εξωτερικής Δράσης, με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προσπαθούμε να συντονίσουμε καλύτερα την πολιτική μας. Προσπαθήσαμε λοιπόν όλοι να μπουν όλα αυτά στον κανονισμό για την πολιτική γειτονία, για το μέσο της πολιτικής γειτονία. Οι προτάσεις αυτές είναι ακόμη σε φάση ολοκλήρωσης της διατύπωσής τους, ενώπιον του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ε, ευρύτερα Ε, ε, μάλλον να συντονίσουμε καλύτερα την ε, οικονομική βοήθεια με τις πολιτικές, να αποτιμούμε καλύτερα την αποδοτικότητα και να υπάρχουν να υπάρχει περισσότερη συμπερίληψη της αρχής αυτής περισσότερο για περισσότερα. Θέλουμε περισσότερη στήριξη του Κοινοβουλίου για μια απλοποίηση του προγραμματισμού και γενικά των διαδικασιών. Θέλουμε επίσης να επικεντρωθούμε σε λιγότερες πρωτοβουλίες και να υπάρξει περισσότερη κατανόηση και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για το πώς θα βοηθηθεί η Ρωσία να περάσει σε μια νέα κατάσταση ως ε, ε, ε λήπτης αναπτυξιακής βοήθειας για να επικεντρωθούμε περισσότερο στις έξι αυτές χώρες. Ε, βεβαίως αν δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε όλες μου τις λεπτομέρειες υπάρχει και το γραπτό κείμενο έκανα μια προσπάθεια να σας δώσω μια σφαιρική συνολική εικόνα των προσπαθειών μας στα πλαίσια της ε, παρούσης ε, δημοσιονομικής περίοδου συνδυασμού των οργάνων όλων επίσης να σας περιγράψω ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις πώς τις αντιμετωπίσαμε μέσω των οργανισμών χρηματοδότησης και πώς όλα αυτά μεταφράζονται στη νέα πρόταση που κάνουμε για το χρηματοδοτικό αυτό μέσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κορνάρο για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση. Να προχωρήσουμε γρήγορα στον δεύτερο μιλητή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Χάινς Όπορς, που είναι διευθυντής ε, των επιχειρήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε καθυστερήσει ένα τέταρτο κατά την έναρξη. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε σύντομοι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα και οι βουλευτές να θέσουν ερωτήσεις στο τέλος. Κύριε Όπερς. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίδεται να παρουσιάσω τις ε, δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επιτρέψτε μου σύντομα να σας θυμίσω τι είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είμαστε η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η οι ε, μέτοχοι λοιπόν είναι τα κράτη-μέλη. Χρηματοδοτούμε προγράμματα για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το κάνουμε με την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε συλλέξει εδώ και πάνω από 50 χρόνια το οποίο σημαίνει ότι δεν εξετάζουμε τα προγράμματα μόνο από την οικονομική πλευρά, όπως κάνουν οι εμπορικές τράπεζες. Δεν επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στην οικονομική ανάλυση, αλλά εξετάζουμε και τις τεχνικές και οικονομικές πτυχές του κάθε προγράμματος, ώστε να φροντίζουμε το πρόγραμμα στο σύνολό του να είναι βιώσιμο και σκόπιμο από τραπεζικής, οικονομικής και τεχνικής άποψης. Στηρίζουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η αξιολόγησή μας ε, λοιπόν ε, εξετάζει και το θέμα των δημοσίων συμβάσεων και περιβαλλοντικά θέματα, ώστε να διασφαλίζουμε κάθε πρόγραμμα που χρηματοδοτούμε να ευθυγραμμίζεται πλήρως με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται από εξωτερικές εντολές και τρεις κατηγορίες έχουμε και ακριβώς ε, θέλω να σας εξηγήσω τι ρόλο παίζει εδώ η γειτονία, η διάσταση της γειτονίας. Ε, έχουμε λοιπόν τις ε, ε χώρες στην πρωταξιακή τους φάση, Κροατία, Τουρκία. Έχουμε την, τις γειτονικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Νότο και την Ανατολή και κατόπιν επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη, στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Ε, αυτά ως μια γενική επισκόπηση. Ε, βλέπετε εδώ στο χάρτη που δραστηριοποιούμαστε στην Ανατολή. Ε, καταρχήν λοιπόν στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ε, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία ε, και Αρμενία. Δεν δραστηριοποιούμαστε στην Λευκορωσία. Ε, εδώ οι δράσεις συντονίζονται με την ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Στο Αζερβαϊτζάν περιμένουμε να δραστηριοποιηθούν πάρα πολύ σύντομα. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των ε, διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία πλαίσιο που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δραστηριοποιηθεί σε μια χώρα. Κοιτάμε ανατολικά, δραστηριοποιούμαστε και στην Ρωσία στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας καθώς και στην Κεντρική Ασία, αυτή τη στιγμή στο Καζακστάν και το Τατζικιστάν. Αν κοιτάξουμε τους στόχους ε, της εντολής μας, επικεντρωνόμαστε καταρχήν σε ε, τοπική ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Στηρίζουμε δηλαδή κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, έχουμε την ανάπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής υποδομής. δρόμους, για παράδειγμα ε, ε, ε, έργα παροχής ύδατος και στον κοινωνικό τομέα προγράμματα εκπαίδευσης. Και τέλος, μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Αυτά καλύπτονται από την εντολή και αποτελούν τις βασικές αρχές που διέπουν τις δραστηριότητές μας. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Θα σας δώσω αργότερα το ε, συνολικό ποσό ανά έτος. Ε, το ε, συνολικό ποσό που καλύπτει εντολή ανέρχεται σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ και η βασική χώρα στην οποία πηγαίνουν τα χρήματα που εξηγείται από το μέγεθος της χώρας είναι η Ουκρανία που λαμβάνει περίπου το 70% των πόρων μας και ακολουθούν η Γεωργία, η Μολδαβία και η Αρμενία. Κατά κεφαλήν η Γεωργία και η Μολδαβία ε, λαμβάνουν ε, μεγαλύτερο ποσοστό στην περιοχή. Αν κοιτάξουμε τους διάφορους τομείς, σε τι ε, χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κυρίως σε μεταφορές και ενέργεια χρηματοδοτεί. Είναι οι κλασικοί τομείς όπως συνήθως ξεκινούν οι δραστηριότητές μας και κατόπιν επεκτείνονται και σε άλλους τομείς. Ε, επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αποτελούν σημαντικό ποσοστό των δικαιούχων, 30% περίπου, και οι κλιματικές δράσεις που ανέφερα νωρίτερα ε, δεν είναι ακριβώς αποκλειστικό κριτήριο επιλεξιμότητας, αλλά φροντίζουμε και στη μεταφορά, για παράδειγμα, στις μεταφορές, ε, να συμμορφωνόμαστε με το ε, σχέδιο για την κλιματική αλλαγή. Εδώ βλέπετε τις δραστηριότητες μας ε, στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για το διάστημα μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, μέχρι το τέλος του 2012. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν ε, δημιουργούμε επαφές επιτόπου και κατόπιν από το 2010 και μετά αναπτύξαμε πλήρως ε, το πρόγραμμά μας. Το 2012 τα ποσά ε, που δόθηκαν στις χώρες ανέρχονται σε 920 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λοιπόν έχει αναπτύξει πλήρως τις δραστηριότητε της ε, και ε, θα μπορέσουμε σίγουρα να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Τι έχουμε μάθει από αυτήν την πρώτη εντολή. Καταρχήν χρειαζόμαστε πολύ στενή σχέση με όλους τους παράγοντες επιτόπου. Την κυβέρνηση, αυτούς που προωθούν ε, τα προγράμματά μας, Και ο λόγος ύπαρξής μας άλλωστε συνδέεται με τις ε, ευρωπαϊκές αποστολές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Φροντίζουμε λοιπόν να στηρίζουμε μόνο προγράμματα ε, στα οποία να εφαρμόζονται οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Η βασική τομή για μας πέρα από την ε, χρηματοδότηση που φυσικά είναι το κύριο έργο μας, αλλά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι καλή προετοιμασία των προγραμμάτων, να φροντίσουμε να τηρούνται οι κατευθυντήρες γραμμές όσον αφορά το περιβάλλον και όσον αφορά τις δημόσιες ε, συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι έτσι συμβάλλουμε στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών. Ο κύριος Κορνάρο. Αναφέρθηκε πριν στον ε, συνδυασμό της τεχνικής βοήθειας ε, και των ε, χρηματοδοτικών δωρεών, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη για επενδύσεις στον τομέα στην περιοχή αυτή, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να στηρίξουμε την εφαρμογή των προγραμμάτων με πόρους αλλά και με τεχνική βοήθεια. Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, όπως σας έδειξα πριν, έχουμε κάνει πολλά στον τομέα μεταφορών και ενέργειας. Και Πιο πρόσφατα, μετά την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση της εντολής, έχουμε αυξήσει τις δραστηριότητές μας στον ιδιωτικό τομέα, ε, χρηματοδοτώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, θα θέλαμε να επικεντρωθούμε και θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα ε, όσον αφορά την στήριξη της εφαρμογής των προγραμμάτων. Δηλαδή, να έχουμε συνδυασμένη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Χρειαζόμαστε στενές θεσμικές σχέσεις, όχι μόνο για την εφαρμογή και χρηματοδότηση των προγραμμάτων, αλλά θέλουμε να μεταφέρουμε τις ευρωπαϊκές αξίες στις χώρες αυτές, θέλουμε να αυξήσουμε την τοπική μας παρουσία και έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε γραφεία στην περιοχή αυτή. Στο Κίεβο ήδη, όχι ακόμα στις άλλες χώρες και στη Μόσχα σύντομα θα έχουμε γραφείο και βέβαια ε, συνεργαζόμαστε στενά με την ε, ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο μέλλον θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στα περιβαλλοντικά προγράμματα και στην εκπαίδευση. Να πω λίγα πράγματα για τη Ρωσία. Η Ρωσία φυσικά δεν συμμετέχει στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, αλλά θεωρούμε την Ρωσία πολύ σημαντική και φυσικά Πρέπει να συνομιλούμε με τους εταίρους αλλά και με τη Ρωσία. Και πάντα σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουμε εντοπίσει τρεις τομείς όπου μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ε, χρηματοδότηση προγραμμάτων ε, στα πλαίσια του προγράμματος ε, για τον εξυγχρονισμό και προγράμματα ενεργειακής απόδοση. Και για το 2013 έχουμε διαθέσει 200 εκατομμύρια για δάνεια προς τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία παρατήρηση για την εντολή και την ε, εγγύηση. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για μας. Θα έχετε παρακολουθήσει την ε, συζήτηση σχετικά με την ε, αξιολόγηση των τραπεζών συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και χαιρόμαστε που μπορέσαμε να διατηρήσουμε την αξιολόγηση ΑΑΑ διότι μας επιτρέπει να βρούμε χρήματα στις κεφάλαια με πολύ ελκυστικούς όρους, ώστε να έχουμε την υψηλότερη δυνατή μόχλευση. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, ποτέ δεν έχει προσφύγει ε, στην ε, εγγύηση, το οποίο από πλευρά προπολογισμού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσο. Και αν κοιτάξουμε πέρα από το τι κάναμε στι χώρε τη Ανατολική Εταιρική Σχέση, το συνολικό διάστημα που ξεπερνάει το διαστημα 2017 2007-2013, ε, μόνο δύο φορέ ε, η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προσφύγει ε, στο μέσο τη εγγύηση. μία φορά για την πρώην Ιουκοσλαβία και μία φορά για την Αργεντινή και όλα τα ποσά επεστράφησαν Είναι λοιπόν πάρα πολύ αποτελεσματικό μέσο όσον αφορά τον προπολογισμό, αλλά και όσον αφορά την διατήρηση τη αξιολόγηση ΑΑΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σα και σας ευχαριστούμε επίσης ε, που ήσασταν σύντομος. Ε, να προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Όλαφ Όσικα, Διευθυντή του Κέντρου Ανατολικών Μελετών στην Πολωνία. Θα μας ε, παρουσιάσει μια κριτική απόψη της διαχείρισης και εφαρμογής των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Και πόσον είπατε ότι θα εκφράσω την άποψή μου για αυτήν την ε, εταιρική σχέση, θα το κάνω. Καταρχήν, θα ήθελα να θυμίσω κάποιους παράγοντες που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν μιλάμε για ε, χρήματα. Δεν είναι μόνο πόσα δαπανώνται, αλλά και πώς δαπανώνται, καθώς επίσης και ποιοι είναι οι ε, φορείς, ε, τα κράτη δηλαδή με τα οποία έχουμε να κάνουμε. Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τη δημιουργία της εταιρικής, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και είναι πολύ νωρί για να προβούμε σε τελικές, τελικά πορίσματα. Αν και είναι καλή καλό το χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να δούμε, να κάνουμε μια αξιολόγηση. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για χώρε που δεν λειτουργούν σε ένα στρατηγικό κενό. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν οι συμφωνίες Σύνδεση, υπάρχει η Ρωσία με την ιδέα της Τελωνιακή Ένωση και άλλα προγράμματα. Καθώς παρακολουθούμε λοιπόν την πολιτική αυτών των χωρών, παρακολουθούμε την κατάσταση καθημερινά, βλέπουμε λοιπόν πως η Ρωσία δεν ε, έχει μεν ε, μέσα γυθνίασης, ωστόσο παρέχει πρόσβαση στις μεγαλύτερες εταιρείες αλλά και στις ε, επιχειρηματικές κοινότητες και τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καν να έχει κάποιο συγκεκριμένο δημοσιονομικό μέσο ή γραμμές. Τρίτον, έχουμε να κάνουμε με έξι πολύ διαφορετικές χώρες. Πολύ διαφορετικές, διαφορετικές φιλοδοξίες, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικοί στόχοι, Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν αξιολογούμε την δαπάνη των ευρωπαϊκών χρημάτων. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός ότι υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Ποιος είναι ο απότερο στόχο τη της ανατολική εταιρική σχέση, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν περιμένουμε να αποδώσουν κάτι αυτές οι χώρες. Μιλάμε για δυνητική μελλοντική προσχώρηση στην Ένωση, για πολιτική συνεργασία, για οικονομική ολοκλήρωση, γιατί από αυτό εξαρτάται τι μπορούμε να έχουμε ως ε, ε, ανταπόδοση από τις χώρες αυτές. Δηλαδή, όταν εμείς δεν ξέρουμε και δεν ξέρουν και οι εταίροι μας ποιος είναι ο απότερος στόχος της ανατολικής ε, εταιρικής σχέσης, πραγματικά είμαι επιφυλακτικός όσον αφορά την αμοιβαιότητα. Όσον αφορά δηλαδή τις βαθιές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα για το μέσο ανατολικής εταιρικής σχέσης πάντοτε είναι πρόβλημα και εκτιμώ το ότι είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πρώτη αυτή εισήγηση με όλα αυτά τα προγράμματα και τα χρήματα που χορηγούνται σε καθένα από αυτά τα προγράμματα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε ακριβώς πόσα χρήματα θα πανάει η Ένωση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Στην αρχή προβλέπονταν 600 εκατομμύρια ευρώ. Ε, από αυτό το μέσο. Τώρα μιλήσατε για 2,8 δις. Πιστεύω πως είναι αυτός ο σωστός αριθμός, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι σαφές και δεν είναι σαφές για τις χώρες εταίρους από πού προέρχονται τα χρήματα. Υπήρχαν διάφορα προγράμματα, ίσως πολλά προγράμματα, δισκορπίζονται τα χρήματα και τελικά αυτό που ακούμε πολλα προγραμματα δυσκορπιζονται τα χρηματα και μιλάμε με τις, ε, συνομιλούμε με τις χώρες εταίρους, ξέρουν πως υπάρχει δημοσιονομική στήριξη, ότι υπάρχει ένα βασικό εργαλείο, ένα βασικό μέσο για την, ε, τα προγράμματα δημιουργίας ε, θεσμών, οικοδόμησης θεσμών, υπάρχει το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών. Ξέρουν ότι υπάρχει μια τεχνική βοήθεια, αλλά αν έπρεπε να πω ας πούμε στους Ουκρανούς συναδέλφους ή στους Γεωργιανούς συναδέλφους ότι 2,8 δι ευρώ υπάρχουν για την ανατολική εταιρική σχέση, φαντάζομαι πως θα εκπλήσονταν, γιατί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα ποσά που τους περιμένουν για να δαπανηθούν στις χώρες τους είναι θέμα μάλλον επικοινωνίας ή θέμα της, του σύνθετου χαρακτήρα της χρηματοδότησης της Ένωσης. Τώρα κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την αντίληψη των εταίρων ε, αυτών για την βοήθεια. Καταρχήν θεωρούν ότι αυτού του είδους η βοήθεια, τεχνική βοήθεια μπορεί να προσφέρει και βράχει πρόθεσμη οικονομική στήριξη, αλλά όχι ως βοήθεια που θα στηρίξει μια βασική μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση με βάση τα ευρωπαϊκά χρήματα. Ε, και αυτό αντικατοπτρίζει αυτή την κατάσταση που αναφέραμε, ότι δηλαδή δεν ξέρουν ποια είναι, αν υπάρχει προοπτική να προσχωρήσουν στην Ένωση ή όχι χρειάζονται τα χρήματα, χρειάζονται διαχείριση, χρειάζονται τεχνική βοήθεια, αλλά στην ουσία δεν συνδέουν τη χρηματοδότηση την ευρωπαϊκή με την αλλαγή ή τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας των χωρών τους. Δεύτερον, μετά από τέσσερα χρόνια φαίνεται πως η ανατολική εταιρική σχέση δεν έχει ε, επηρεάσει πολιτικά τουλάχιστον όχι, ε, δεν, έχει, δεν έχουν υπάρξει απτές, ε, απτά αποτελέσματα η επιπτώσεις. Δεν, δεν έχει φτάσει στον απλό πολίτη. Δεν ξέρουν καν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ρόλο στη ζωή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στους απλούς πολίτες της Ουκρανίας, της Μολδόβα και της ε, Γεωργίας δεν υπάρχει. Δεν το λαμβάνουν υπόψη δηλαδή ως παράγοντα. Ίσως το πρόβλημα να είναι η έλλειψη όχι έλλειψη, αλλά εν πάση περιπτώσει η λιγοστή επιρροή μπορεί να εξηγείται και από το γεγονός ότι αυτό που λείπει είναι ένας μηχανισμός για θετικούς όρους, αυτό που λέγαμε θετικές προϋποθέσεις, το more for more. Περισσότερος κόσμος όταν μιλάμε για, με διοικητικούς υπαλλήλους των χωρών αυτών λένε ανοιχτά πως δεν έχουν κανένα κίνητρο να μπλακούν περισσότερο γιατί άσχετα από την πρόοδο τα χρήματα τους έχουν δοθεί εκ των προτέρων τα περισσότερα ούτως ή άλλως. Πιστεύουν δηλαδή πως ε, κάποια χρήματα υπάρχουν, μπορεί να μην είναι και ε, τεράστια ποσά, ε, πάντως θα τα πάρουν ούτως ή άλλως. Δεν έχουν κίνητρο να δουλέψουν περισσότερο προσωπικά, ούτε και η διοίκησή τους έχει κίνητρο. Αυτό είναι σημαντικό ίσως να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση περισσότερα για περισσότερα, more for more, γιατί έτσι ίσως να υπάρξουν αντιδράσεις για, τις, για αλλαγές. Και όταν σκεφτούμε την περιοχή, τις χώρες της Ανατολικής ε, Τερκής Σχέσης, βλέπεις πως ε, οι κοινωνικές, οι πολιτικές αλλαγές μπορούν να γίνουν και μία ανοιχτή κάποιες φορές. Χρειάζονται λοιπόν μέσα για να ανταμείβονται αυτοί που θέλουν περισσότερα, που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις της χώρας τους. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το, το μέσο και κατά κάποιο τρόπο παγιώνεται η κατάσταση στις χώρες αυτές. Αυτές που προχωρούν, προχωρούν ούτως ή άλλως, αν και θα μπορούσαν να προχωρήσουν και περισσότερο, αυτές που διαφορούν συνεχίζουν να διαφορούν. Δεν κάνουν κάτι παραπάνω γιατί τα χρήματα θα υπάρχουν ούτως ή άλλως. Τέλος, υπάρχει πρόβλημα που αναφέρετε και εσείς στην δική σας εισήγηση για το ποιον πρέπει να προσεγγίσουμε. Φαίνεται πως η Κομισιόν έχει περιοριστεί στη συνεργασία της με τη κυβέρνηση και τους διοικητικού μηχανισμούς των χωρών εταίρων. Όμως χρειάζεται να φτάσουμε στους απλούς πολίτες, όχι μόνο στην κοινωνία των πολιτών, της ΜΚΟ, γιατί και αυτό είναι τμήμα του προβλήματος ότι δηλαδή υπάρχει μια μικιοκρατία, δηλαδή θεσμοί που είναι υπέρ της Ευρώπης, ξέρουν πώς να αναζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση, δεν έχουν με τον απλό κόσμο στις περιοχές της Υπέθρου, στην ε, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. αν υπάρχει. Και πρέπει να μπούμε δηλαδή βαθύτερα στην κοινωνία για να υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα και να υπάρξει κάποια διαφορά. Είναι αόρατη η χρηματοδότηση της Ένωσης για τον απλό κόσμο. Υπάρχει, είναι ορατή για του δημόσιους οργανισμούς και τις δημόσιες διοικήσεις, αλλά αν κατέβεις παρακάτω η Ένωση δεν υπάρχει. Ως μια οντότητα που μπορεί να δώσει χρήματα και να κάνει καλά πράγματα για τον απλό κόσμο. Κλείνοντας, μετά από τέσσερα χρόνια βλέπουμε λοιπόν πως οι πολιτικές και οι κοινωνικές συνθήκες σε όλες τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης δεν έχουν, αν δεν έχουν επιδεινωθεί έχουν μείνει στάσιμες. Η Ουκρανία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Η Ουκρανία στην Ουκρανία η πολιτική και η κοινωνική κατάσταση επιδεινώνεται, η Γεωργία είναι ένα ερωτηματικό, η Μολδόβα αγωνίζεται, αλλά βλέπουμε πως μετά από την κατάρρευση της κυβέρνησης, λίγους μήνες πριν από τη διάσκεψη κορφής του Βίλνιους, κινδυνεύει να χάσει τη στιγμή, τη στιγμή την κατάλληλη που με τις πιο φιλόδοξες χώρες όπως είναι η Μολδόβα, η Γεωργία ε, και η Ουκρανία κατά περιόδους. Αυτό που χρειάζεται είναι λιγότερα μέσα, αλλά με σαφείς προτεραιότητες. Αν ορίζουμε ότι οι πολιτικές ελίτ κάποια χώρα δεν ενδιαφέρονται να μπουν στην Ένωση, θα πρέπει τότε η προτεραιότητα να είναι η κοινωνία, οι νέοι, να φτάσουμε δηλαδή σε, αυτό, σε αυτές τις ομάδες. Δεύτερον, απλοποίηση των διαδικασιών. Όσο πιο περίπλοκα είναι τα προγράμματα, τόσο λιγότερο προσιτά είναι όχι μόνο για τους ε, διοικητικούς μηχανισμούς, αλλά και για τις διάφορες ομάδες, ε, μη κυβερνητικέ κτλ. Τέλος, αυτό που θα πω τελειώνοντας είναι ότι θα πρέπει με καλύτερο τρόπο να εξηγήσουμε πόσα χρήματα υπάρχουν δυνητικά ε, τα νούμερα είναι αδιαφανή. Κανένας δεν πρόκειται να πιστέψει πως υπάρχουν τουλάχιστον 3 δις ευρώ που τους περιμένουν από, αυτούς, τους, ε, από αυτές τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Αυτό δεν το έχουμε εξηγήσει ε, και αν δεν το καταφέρουμε να το εξηγήσουμε εμείς θα συγκρινόμαστε, ούτως ή άλλως συγκρινόμεθα από τους επιχειρηματικούς ε, κύκλους, από το διοικητικό μηχανισμό των χωρών αυτών με τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι παρούσα. Τα ρωσικά εξάλλου είναι η γλώσσα, η κοινή όλων αυτών των χωρών. Πολιτιστικά και άμεσα η Ρωσία είναι λοιπόν πολύ παρούσα, εμείς όχι. Αν και δίνουμε πολλά χρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Uh, for that present... Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Ε, συνοπτική. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Να περάσουμε τώρα στην κυρία Γιολάντα Ταζάνκα που είναι το Ίδρυμα για Ευρωπαϊκές Σπουδές ε, και το Πανεπιστημίο του Woods Lodge. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Ιολάντα Ταντέσκα. Ευχαριστώ που μου δώσατε δυνατότητα να μιλήσω σε ένα τόσο διακεκριμένο ακροατήριο. Έχω ε, ασχοληθεί με αυτήν την ε, εταιρική σχέση Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, έχει κάνει η Ένωση μεγάλες προσπάθειες για να βοηθήσει την ευρωπαϊκή ενοποίηση και να υποστηρίξει τη διαδικασία νομικής εναρμόνισης. Και τα θέματα αυτά είναι πάντα επίκαιρα. Χαίρομαι λοιπόν που είμαι παρούσα για να μοιραστώ με σας μερικές σκέψεις για τα θέματα αυτά. Εδώ και δέκα χρόνια εργάζομαι σε μία από αυτές τις χώρες. Οι συνεργάτες μου και εγώ αναλάβαμε ένα περίπλοκο και πολύ ευρύ καθήκον. Να ενισχύσουμε τη δυνατότητα λειτουργίας του κράτους, ούτως ώστε να προσεγγίσει τα ενωσιακά πρότυπα. ιδιαίτερα στον τομέα προσαρμογής της νομοθεσίας και τη θεσμική και διοικητική βελτίωση της λειτουργίας. Βεβαίως σήμερα θα κυρίως με την ε, εξέβρεση του καλύτερου τρόπου λειτουργίας χορήγησης ε, ενωσιακών χρηματοδοτήσεων εντός αυτής της ε, πρωτοβουλίας ανατολικής εταιρικής σχέσης. Αλλά διτά πρέπει να δούμε το θέμα αυτό. Δηλαδή, από τη μία από την ε, προοπτική συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων και από την προοπτική της πρακτικής εφαρμογής όσων αποφασίζουν οι εταίροι. έχοντας παρατηρήσει πώς λειτουργούν ε, όλα αυτά τα πράγματα, θα σας εξηγήσω την άποψή μου και θα κάνω συστάσεις και προς την ε, πλευρά που χρηματοδοτεί και προς τους παραλήπτες της χρηματοδότησης, των χρηματοδοτήσεων. Τρία είναι τα σημεία κλειδιά Λοιπόν, τρία είναι. Ε, έλεγχος, μεθοδολογία και βιωσιμότητα. Θα μπορούσα να τα στείλω σε ένα SMS στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα, επειδή η τεχνική βοήθεια προσπαθεί να εφαρμόσει συγκεκριμένες πλευρές του, κοινοτικού κεκτημένου βοηθάει δίνοντας μια ε, θεωρητική πλευρά στην ε, τεχνική βοήθεια για να ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητες και να δημιουργήσει πολύ πιο σταθερές, ε, σταθερούς θεσμούς. Για να είναι αποτελεσματική η τεχνική βοήθεια πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του παραλήπτη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί η κάθε πρωτοβουλία να έχει αποτελέσματα και να παίξει ζωτικό ρόλο στις διαδικασίες ε, μεταβολών στις ε, ωφελούμενες χώρες. Η τεχνική βοήθεια όμως πρέπει να βασίζεται και στην συνένεση από την πλευρά των ωφελουμένων. Δηλαδή πρέπει και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν στις διαδικασίες. Δηλαδή η Ένωση βοηθάει την ε, εφαρμογή των ε, μεταρρυθμίσεων και η χώρα που λαμβάνει την ενίσχυση δεσμεύεται να κάνει αυτές τις αλλαγές. Για να είναι αποτελεσματική πλήρως λοιπόν κάθε μέσο τεχνικής βοήθειας πρέπει να βασίζεται σε δύο συνθήκες. Πρώτον, Πρέπει να έχει καλώς καθορισμένο στόχο και σκόπιμο. Και από τις δύο πλευρές. Και δεύτερον, η ανατολική γειτονία και συγκεκριμένα οι δημόσιοι φορείς των χωρών γειτονίας που είναι ε, που, των χωρών λοιπόν γειτονίας πρέπει να καθορίζουν σαφώς ποιος οργανισμός θα εφαρμόσει τη συγκεκριμένη δράση. η μεταγραφή των ε, κοινοτικών προδιαγραφών στο εθνικό ε, νομοθετικό πλαίσιο προκαλεί προστιθέμενη αξία στον παραλήπτη. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Εγώ διαπίστωσα ότι πολλοί δημόσιοι πάλι στις χώρες αυτές είναι καλώς καταρτισμένοι, μιλάνε γλώσσες, έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση. Άρα η τεχνική βοήθεια πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένης φύσης. θα πρέπει να εδρεώσουν στις ε, μεθόδους διακυβέρνησης των χωρών αυτών τις ενωσιακές μεθόδους. Στην καθημερινή εργασία των ε, ε, διοικήσεων στις χώρες αυτές. Και είμαστε στην σωστή συγκυρία για να σκεφτούμε και τι είναι πλευρές μπορεί να λάβει η τεχνική βοήθεια λόγω των ε, συμφωνιών σύνδεσης. Η τεχνική λοιπόν βοήθεια είναι σε μια εκπληκτική κατάσταση. όσον αφορά την άποψη, την ε, θεώρηση των αντιπροσωπιών της Ένωσης στις χώρες αυτές για το πώς δηλαδή βοηθάνε τις χώρες αυτές. Ορισμένες αντιπροσωπείες είναι απόλυτα αντίθετες προς τις προσπάθειες που κάνουν οι ομάδες προγραμμάτων, τις διαπραγματεύσεις, την προπαρασκευή των διαπραγματεύσεων. Ορισμένες αντιπροσωπείες, από την άλλη μεριά, βοηθάνε και έχουν πολύ καλή θέληση. Ένας από τους ε, κύριους στόχους τεχνικής βοήθειας είναι να πείσει τους παραλήπτες, τις χώρες αυτές, ότι η πολιτική ευρωπαϊκής ενοποίησης πρέπει να θεωρηθεί εσωτερική και όχι εξωτερική πολιτική από πλευράς τους. Διότι στις συμφωνίες ε, σύνδεσης προβλέπονται νέες νομικές δεσμεύσεις. Πρέπει να υπάρχει μια συστημική και περίπλοκη, λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ήδη μια συστημική και πλήρης προσέγγιση για την μεταγραφή του ευρωπαϊκού δικαίου και την προσαρμογή στην ενωσιακή και ε, διεθνή πραγματικότητα και δεσμεύσεις των χωρών αυτών η προσαρμογή των νομοθετημάτων θα είναι το κύριο όργανο Η νομική λοιπόν αυτή προσαρμογή σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια ε, ευρεία αναθεώρηση και να υπάρχει μια σαφής θεσμική βάση και να υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες και σε νομοθετικό και σε εφαρμοστικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα νέο πρότυπο για τη διαδικασία νομικής προσέγγισης και προσαρμογής μέσω συντονισμένης μεθοδολογίας. Λοιπόν, τα κράτη αυτής της περιοχής θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οπότε, πρέπει να αυξηθούν οι ικανότητες των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν αναλάβει τα καθήκοντα προσαρμογής στο ενωσιακό και εκτιμένο. Η τεχνική βοήθεια βεβαίως θα τους υποστηρίξει, θα τους καταρτήσει. και θα καταρτήσει και τους εκπαιδευτές. Επίσης, οι ενωσιακές ενισχύσεις πρέπει να στοχεύουν και στην ενημέρωση των εθνικών βουλευτών. Τους ε, παραμελούμε, ούτως ώστε να έχουν το κατάλληλο προσωπικό Επίσης να βοηθήσουμε άλλες επαγγελματικέ ομάδες, πανεπιστημιακούς, τους δικαστές, τους μεταφραστές. Μέχρι το 2012, τονίζω, το πρόγραμμα για το οποίο είχα την ευθύνη ήταν το μόνο ενωσιακά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας που εργαζόταν στην ε, Ουκρανία ενώ υπάρχουν ε, πολύ ενεργοί ε, οργανισμοί από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η τεχνική βοήθεια παίζει επίσης πολύ βασικό ρόλο, όπως είπα ήδη. Παίζει ρόλο για να δημιουργήσει κέντρα ενημέρωσης, ε, πλατφόρμες ενημέρωσης για την ε, διάδοση ε, ενημέρωση για την Ένωση και την διεξαγωγή εκστρατιών ενημέρωσης. Η δική μου λοιπόν ομάδα μαζί με αμερικανικούς φορείς έχουν δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ενημέρωσης και Με βάση την απόφαση τη ε, ενωσιακή αντιπροσωπεία εκεί, τελικά την ευθύνη λειτουργία την ανέλαβε ο φορέα των Πολιτειών. Η τεχνική βοήθεια πρέπει επίσης να βοηθήσει να δημιουργηθούν, να δημιουργηθούν, να δημιουργηθούν θύλακοι εμπειρογνωμόνων πολύ ψηλού επίπεδου. Διότι μία ιδιαιτερότητα της περιοχής είναι ότι τη μερίδα του λέοντος ε, την εργασία την κάνουν οι εγχώροι εμπειρογνώμονες αλλά οι δικοί μας εμπειρογνώμονες παίζουν επικουρικό ρόλο. Έτσι έχουν την ευθύνη οι τοπικοί εμπειρογνώμονες για να αξιοποιήσουν αυτά που μαθαίνουν με τη βοήθεια κάποιων Ευρωπαίων, δηλαδή ενωσιακών ε, συμπαραστατών. Υπάρχουν λοιπόν έμπειροι εμπειρογνώμονες που τους ε, αναγνωρίζουν και τους σέβονται οι εγχώροι εμπειρογνώμονες και που έχουν ήδη βοηθήσει. Επιπλέον, η ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να συμβάλλει για να προωθηθούν ευρείας κλίμακος ε, διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα η κοινοβουλευτική συνέλευση Euronest, που είναι μια θαυμάσια πλατφόρμα, ένα θαυμάσιο βήμα δια κοινοβουλευτικής ε, συζήτησης μεταξύ των χωρών της Ένωσης και των χωρών της περιοχής και το Corla που είναι ε, φορές συνεργασίας ε, των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ποια είναι η άποψή μας ε, ημών που εφαρμόζουμε τεχνική βοήθεια. Γιατί πρέπει και εμείς να κάνουμε πολλές περαιτέρω προσπάθειες Πρέπει να βοηθήσουμε κάθε νομική και ε, προσπάθεια διαμόρφωσης πολιτικής στην περιοχή αυτή. Πρέπει να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση και να αντιλαμβανόμεθα τις διαφορετικές ε, πλευρές της πολύπλοκης τοπικής πραγματικότητας. Πρέπει να βοηθούμε την περιφερειακή συνεργασία της Ένωσης γενικότερα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο την εμπιστεύονται οι τοπικοί εταίροι. Η καθημερινή συνεργασία πρέπει να αφορά όλους τους κύριους φορείς και να εντάσσεται η εργασία μας ε, στις προσπάθειες ε, όλων των άλλων που συμμετέχουν. Για παράδειγμα, η διδημοποίηση, το ΣΥΓΜΑ, το ΤΑΙΕΞ, και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Στρατηγική κάθε προσπάθειας τεχνικής βοήθειας. Δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε στην χορήγηση των όσων έχουν συμφωνηθεί. Κυρίως βοήθεια σημαίνει απτά αποτελέσματα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, κάθε καθήκον που αναλαμβάνει μια ομάδα τεχνικής βοήθειας πρέπει να ε, αναλαμβάνεται ε, σε τρεις φάσεις. Πρώτα απ' όλα προκατακτικές συναντήσεις, ταυτοποίηση δηλαδή των στόχων και εξοικείωση με το τοπικό περιβάλλον, εφαρμογή και μετά βοήθεια μετά την εφαρμογή, εκ των υστέρων. Ποιες αδυναμίες διαπιστώσαμε στην εργασία μας. Πρώτα απ' όλα, έλλειψη εδραίωσης της λεγόμενης θεσμικής μνήμης, δηλαδή της κληρονομίας κάθε προγράμματος. Τι αφήνει πίσω. Μόλις ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα, είναι σαν ε, να μην είχε γίνει ποτέ. Δεν μπορούν ε, κατόπιν προγράμματα να αποφεληθούν από την πείρα που ε, συνελέγει κατά την εφαρμογή ενός προγράμματος. Άλλη αδυναμία. Δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπιών της Ένωσης και των ομάδων τεχνικής βοήθειας. Ορισμένες φορές ε, δεν υπάρχουν καθόλου επαφές, σε άλλες περιπτώσεις απλώς δεν είναι τακτικές. Οι ομάδες τεχνικής βοήθειας θέλουν και αυτές κάποια βοήθεια από τις αντιπροσωπείες. Επιπλέον, δεν ε, εξετάζονται αρκετά τα αποτελέσματα της τεχνικής βοήθειας, δεν αναγνωρίζονται. Μας δημιουργείται η εντύπωση ότι οι αρμόδιες τη Ένωση της δεν διαβάζουν καν τις εκθέσει μα. Δεν υπάρχει συστημική συνέχεια. Οπότε έχουμε ασυνέπειες και έλλειψη συστηματικότητας. Και τέλος, οι ενωσιακές χρηματοδοτήσεις ε, αντιμετωπίζονται ως τυχαίες, ότι δεν εντάσσονται σε ένα ε, συστηματικό πλαίσιο. Συστάσεις τώρα. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει σταδιακή βελτίωση της τεχνικής βοήθειας που πρέπει να είναι σαφής και να γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αλλά όχι ιδιαίτερα απαιτητικά. Απαιτητικά βεβαίως, αλλά όχι υπερβολικά. Πρέπει να υπάρξει εκλέπτυνση και ενίσχυση της συνεργασίας με τις αντιπροσωπείες και τους ε, παραλήπτες της βοήθειας. Πρέπει να υπάρχει καθημερινή επαφή μεταξύ των αντιπροσωπιών και των ομάδων τεχνικής βοήθειας. Και θα πρέπει να δημιουργήσουμε δομές ε, συντονισμού με εκπροσώπους της Ένωσης, εκπροσώπους άλλων ε, χορηγών και τις ομάδες τεχνικής βοήθειας για να ανταλλάσσουν απόψεις, να συζητάνε τις εξελίξεις, να δρουν συντονισμένα και να εκπονούν κατευθυντήρες γραμμές για τα επόμενα προγράμματα. Και υπάρχουν τέτοιες δομές, υπήρξαν σε ορισμένες φάσεις και κατόπιν διαλύθηκαν. Ναι, ναι, τελειώνω, τελειώνω. Τώρα, για να εποφεληθούμε από την στήριξη των διεθνών εμπειρογνωμόνων, πρέπει να δημιουργήσουμε θυλάκους τέτοιων ε, εμπειρογνωμόνων ειδικού επίπεδου που να συνοδεύονται από υψηλού επίπεδου ε, τοπικούς δημοσίους υπαλλήλου για να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία και να αποφύγουμε λανθασμένες συμβουλές. Να αποφύγουμε την έλλειψη συνέχεια στην εργασία μας. οι εκπρόσωποι της Ουκρανικής κυβέρνησης συχνά μου είπαν ότι έχουμε πολύ καλού επίπεδου εμπειρογνώμονες αλλά οι συμβουλές τους είναι υπερβολικά θεωρητικές, αφηρημένες. Δεν μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, μας λένε. Δεν είναι εφαρμόσιμες. Επίσης θα πρότεινα να υπάρξει και ένας μηχανισμός διακρατικής συνεργασίας. Ίσως μια, ένας κοινό ε, τεχνικός οργανισμός ή φορέας για όλη την περιοχή. Σας ευχαριστώ ε, και ευχαριστώ να απαντήσω στις, ε, στις ερωτήσεις σας και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Θα ήθελα να προχωρήσω γρήγορα στους, επόμενους, στους τελευταίους δύο μιλητές μας. Ε, η επόμενη ομιλήτρια ε, θα μας μιλήσει για την, ε, για την πλευρά των μη κυβερνητικών οργανώσεων, Ανά Κριστίνα Λίνκ από το Ίδρυμα Κόνρα Άντεναουερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που καλέσατε το Ίδρυμα Κόνραντ Ατενάουερ να σας μιλήσουμε για τις εμπειρίες μας. Λίγα λόγια για το ίδιο το Ίδρυμα. Για να γνωρίζετε τι είδους οργάνωση είμαστε. Είμαστε ε, ένα γερμανικό πολιτικό ίδρυμα που χρηματοδοτείται από ε, τον Ομοσπονδιακό Προλογισμό της Γερμανίας. Ε, έχουμε 16 εκπαιδευτικές ακαδημίες και από το 1962 και μετά έχουμε διεθνή προγράμματα συνεργασίας μέσω 80 γραφείων σε 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πολυετή προγράμματα συνεργασίας και συνεργαζόμαστε με θεσμικούς εταίρους στις χώρες. Έχουμε τοπικά γραφεία στην περιφέρεια της Ανατολικής Έχουμε ένα γραφείο στην Ουκρανία, ένα στη Μολδαβία. Ε, ε, έχουμε ένα γραφείο στη Λιθουανία που καλύπτει την ε, Λευκορωσία και έχουμε ε, ε, δραστηριοποιούμαστε και στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Ε, και έχουμε και ετήσιο προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2005 και μετά ε, ασχολούμαστε με αιτήσει ε, προς ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση και ακριβώς γι' αυτό μου ζητήθηκε να σας περιγράψω τις εμπειρίες μας. Η δομή της παρουσίασης αυτής είναι αρκετά πρακτική. Θα αναφερθώ λοιπόν σε κάποια προγράμματα που έχουμε στην περιοχή. Επίσης θα σας μιλήσω για τις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές από τη δική μας πλευρά και θα προσπαθήσω να σας, να συγκρίνω την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλων δωρητών. Έχουμε λοιπόν προγράμματα στην περιφέρεια της ε, Ανατολικής Εταιρικής ε, Σχέσης. Ε, θέλουμε να αυξήσουμε την λογοδοσία και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αναφέρθηκε στην αρχή της συνάντησης όπου Είμαστε ένας από τους ε, βασικούς δικαιούχους ε, από πλευράς της κοινωνίας των πολιτών. Ε, είναι λοιπόν ένα έργο 3,4 εκατομμυρίων ευρώ ε, και παρέχουμε υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι ε, πολύ διαφορετικό από αυτό που γίνεται συνήθως. Είμαστε όμιλος εννέα εταίρων, 7 ε, είναι τοπικοί, τοπικές με κυβερνητικές οργανώσεις και ο στόχος του είναι να ενισχύσει το δυναμικό στις οργανώσεις της κοινοτήρας των πολιτών και να βελτιώσει την συνεισφορά του τους. Θα έχουμε δραστηριότητες χαρτογράφηση, οικοδόμηση δυναμικού, στήριξη ad hoc. Ε, επίσης, ε, διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους ε, και ορατότητα του μέσου για την πολιτική γειτονίας, ανατολική πολιτική γειτονίας. Επίσης, έχουμε και κάποιες άλλες συμβάσεις στον νότιο ε, Κάφκασο. Ε, ο προπολογισμό ε, ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια που συγχρηματοδοτείται από το AIDHR. 77% είναι ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση και το υπόλοιπο παρέχεται από το Ίδρυμα Conrad Adenauer. Συμμετέχουν δύο, ευρωπαϊκοί, δύο ευρωπαϊκές και τρεις τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο στόχο είναι να δημιουργηθεί ένα μηχανισμό για τη συνεχή προώθηση τη πολιτική συμμετοχή νέων από ε, γεωργικέ περιοχέ και περιοχέ ε, μειονοτήτων στην Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και Γεωργία, στην κοινωνία των πολιτών ε, και πολιτικές δραστηριότητες στις διάφορες χώρες. Έχουμε διάφορες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ε, την ε, ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτικού υλικού. Έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα μέσα στην οποία οι διάφοροι δάσκαλοι μπορεί να έχουν ανταλλαγέ όσον αφορά την πολιτική εκπαίδευση και έχουμε δημιουργήσει την Ένωση Δάσκαλοι από τον Νότιο Κάφκασο για την πολιτική εκπαίδευση. Επίση, έχουμε παιχνίδια προσωμείωση, το Κοινοβούλιο των Νέων και ε, επίσης έχουμε αυτή την εβδομάδα ε, μια ομάδα ε, φοιτητών που επισκέφτεται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το τρίτο πρόγραμμα λαμβάνει η χώρα στη Λευκορωσία. Δεν μπορώ να σας πω πολλά γι' αυτό επειδή ακόμα πραγματοποιείται και αν σας πω πολλά μπορεί τελικά να ε, την εφαρμογή του και γι' αυτό λίγα λόγια χρηματοδοτείται στα πλαίσια του NSA και ένα αποτελέσματα είναι να δημιουργηθεί ένας ε, μηχανισμός ε, μεταξύ ε, μη κρατικών παραγόντων και τοπικών αρχών στην περιοχή αυτή μέσα από εκπαίδευση, διαβουλεύσεις, παρουσιάσεις, ταξίδια, σεμινάρια κλπ. Αυτά για να σας δώσω μια ιδέα του τι είδου προγράμματα εφαρμόζουμε και θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειε όσον αφορά τις εμπειρίες μας ε, στα διάφορα στάδια ε, υποβολή αιτήσεων και εφαρμογή των προγραμμάτων. Να ξεκινήσω λοιπόν από ε, το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Είναι διαφορετικού τύπου σύμβαση από τα άλλα δύο προγράμματα. Η πρόβλεψη δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2011. Σχετικό ανακοινωθέν δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2012 και αυτό το έγγραφο ε, μιλούσε για την ε, απέτηση να έχουμε τουλάχιστον έναν μη κρατικό παράγοντα από τις ε, χώρες της πολιτικής γειτονίας. Έτσι λοιπόν ήταν αρκετά διαφορετικά αυτά από αυτά που περιμέναμε όταν είδαμε την πρώτη ανακοίνωση τον Οκτώβριο του 2011. Είχαμε μία εβδομάδα για να υποβάλουμε δήλωση μια αίτηση για δήλωση ενδιαφέροντο ε, και τον Οκτώβριο του 2012 με μία 6 εβδομάδε μέχρι τον Νοέμβριο δηλαδή έπρεπε να αναπτύξουμε τη μεθοδολογία μα ε, και ε, να υποβάλουμε όλα τα διοικητικά έγγραφα. Η σύμβαση υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2012, λίγο πάνω από ένα χρόνο δηλαδή κράτησε η όλη διαδικασία. Οι προκλήσεις για μας ήταν οι εξής. Καταρχήν έπρεπε να συμμετέχουν στον όμιλο μη κυβερνητικέ οργανώσει. Αυτό είναι δύσκολο διότι ε, συνήθως οι διαγωνισμοί ε, ε, γίνονται για, για λόγους κέρδους και έτσι λοιπόν ήταν λίγο διαφορετική κατάσταση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το, η άλλη δυσκολία ήταν ότι θα πρέπει να είναι κατοχωρημένοι νομικά στις χώρες αυτές. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες, η Λευκορωσία για παράδειγμα. γενικά λάβαμε 11 δηλώσεις ενδιαφέροντος από τοπικούς οργανισμούς και έπρεπε να έχουμε από κάθε χώρα μια μη κυβερνητική οργάνωση. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει αυτέ όμω δεν καταλαβαίναν ε, τι ακριβώ γινόταν. Και κατά την ε, ε, δήλωση ενδιαφέροντο, δεν ήξεραν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, δεν ήταν πολύ σαφή ο ρόλο του και δεν μπορούσαμε να του εξηγήσουμε τι θα, έπρεπε να τι θα χρειαζόταν να κάνουν αργότερα κατά την εφαρμογή του προγράμματο. Γενικά υπήρχαν αρκετά τεχνικά κριτήρια ε, ε, επιλογής. Έπρεπε να έχουμε τρία ε, διεθνή έργα. Το 50% έπρεπε να εφαρμόζεται από φορείς στην κοινωνία των πολιτών και όλα αυτά θα έπρεπε να είναι από το 2009 μέχρι το 2012. Ήταν αρκετά περιοριστικά όλα αυτά. Δεν υπήρχαν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που να πληρούν τα κριτήρια αυτά. Στην ε, φάση του διαγωνισμού έπρεπε να υποβάλουμε και δικαιολογητικά ε, που είχαν να κάνουν με τα κριτήρια αποκλεισμού, διότι έπρεπε να υποβάλουμε έγγραφα τα οποία δείχνουν ότι δεν ε, έχουμε χρεοκοπήσει, ότι πληρώνουμε τους φόρους μας και ότι δεν έχουμε κάνει διάφορες παραβάσεις. Έγγραφα τα οποία συνήθως δεν αφορούν τους μη κυβερνητικού οργανισμούς, διότι δεν είναι εμπορικοί οργανισμοί. Αυτό λοιπόν δημιούργησε πολλές δυσκολίες σε κάποιες χώρες Τη ε, της εταιρικής σχέσης. Και προς το τέλος, όταν είχαμε υποβάλει την ε, προσφορά μας, ε, λάβαμε κάποιες διευκρινήσει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είχαμε όμως πολύ λίγο χρόνο αντίδραση. Η αρχική προθεσμή ήταν 48 ώρες, ε, όλα έγιναν με φάξ ε, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο πάντα να φροντίζουμε οι ε, απαντήσεις να αποστέλλονται εγκαίρως, διότι ποτέ δεν γνωρίζει κανείς αν οι εταίροι μας είναι διαθέσιμοι εντός αυτού του 24ωρου για να υπογράψουν άλλο ένα έγγραφο ή για να λάβουν διευκρινήσεις από τις δικές τους διοικήσεις. Όσον αφορά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, είχαμε το πρόγραμμα για τον Κάφκασο ξεκίνησε το 2008 με προθεσμία υποβολής ε, το 2008. Ε, ε, το αρχικό έγγραφο ήταν πέντε σελίδων και έπρεπε να περιέχει και μια σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων. Τον Φεβρουάριο του 2009 έπρεπε να υποβάλουμε το σύνολο της αίτησης 31 σελίδες με πολλές λεπτομέρειες ε, σχετικά με τη βιωσιμότητα και άλλε πτυχέ ε, του προγράμματο και τελικά έπρεπε να υποβάλουμε και τον προπολογισμό. Ε, η επιλογή ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2009 και η σύμβαση υπεγράφει τον Οκτώβριο του 2009. Λίγο πάνω από ένα χρόνο κράτησε η διαδικασία αυτή, κατανοητό, διότι ε, ε, μπορούσαν να συμμετάσχουν και μη κυβερνητικέ οργανώσει και η αξιολόγηση απαιτούσε περισσότερο χρόνο. Όσον αφορά το πρόγραμμα για τη Λευκορωσία, ε, ξεκίνησε η διαδικασία τον Ιούλιο του 2011, ε, το αρχικό έγγραφο ε, δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, όπως και η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων ε, και η πλήρη ε, αίτηση υπευλήθηκε τον Νοέμβριο. Η ανακοίνωση σχετικά με την επιλογή έγινε τον ε, Μάρτιο του 2012. Για κάποιο λόγο κράτησε πάρα πολύ μέχρι να υπογράψουμε τη σύμβαση. Τελικά υπεγράφει δηλαδή τον Ιούλιο του 2012 με την αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κίεβο, διότι δεν υπήρχε ακόμα την προσωπία στην Λευκορωσία. Κράτησε λοιπόν αρκετά αυτή η διαδικασία αυτή. Μπορεί όμω αυτό να έχει να κάνει με το γεγονό ότι πρόκειτο για τη Λευκορωσία που είναι η περίπτωση. Όσον αφορά τις προκλήσεις στην ε, διαδικασία υποβολής αιτήσεων ε, ε, και τα στοιχεία αυτά δεν βασίζονται μόνο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Υπάρχει λοιπόν η καταχώρηση Παντόρ, η οποία είναι υποχρεωτική και κάθε οργάνωση θα πρέπει ε, να δώσει το καταστατικό της, ε, της εκθέσεις των ελεγκτών ε, κλπ. Αυτό κρατάει πάρα πολύ καιρό, για, αυτό απαιτεί πάρα πολύ χρόνο για τις τοπικές οργανώσεις, δεν έχουν πάντα έτοιμα τα έγγραφα και μερικές φορές δεν γνωρίζουν τι απαιτείται από αυτούς. δεν υπάρχουν τα πεδία για να ανεβάσει κανείς τα απαραίτητα έγγραφα. Έπρεπε λοιπόν να επισυνευτεί στα άλλα έγγραφα, ε, έπρεπε κάποια έγγραφα να επισυνευτούν σε άλλα. Ο χρόνο αντίδραση ε, ε, ήταν μακρύ σε μερικέ περιπτώσει. Σε κάποιε περιπτώσει έπρεπε να περιμένουμε κάποιου μήνε για να λάβουμε απάντηση και πολύ συχνά λαμβάνει κανείς απλά ένα απόσπασμα από τον οδηγό Παντόρ που συνήθως έχει διαβάσει κανείς προτού να αποστείλει την ερώτηση. Δεν υπάρχει ενιαία γλώσσα για την υποβολή των αιτήσεων. Έχουμε ανεβάσει λοιπόν τώρα το καταστατικό μας ε, σε πολλές γλώσσες τώρα πια, διότι κάθε αντιπροσωπεία ε, ζητάει ε, η αίτηση να υποβάλλεται στη γλώσσα της και υπάρχουν κάποιες επιπλέον απαιτήσει για τα έγγραφα. Όταν υπάρχει όταν θέλουμε να ε, ενισχύσουμε ένα δίκτυο πρέπει να ανεβάσουμε το καταστατικό στο δίκτυο. Ε, ε, υπήρχαν λοιπόν αρκετές δυσκολίε, τι οποίε όμω ξεπεράσαμε. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία υποβολή αιτήσεων για όλε τι γενικέ διευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι περισσότερε φορέ επικοινωνούμε με την Γενική Διευθύνση ΤΕΦΚΟ. Εκεί είναι εναρμονισμένα τα πράγματα, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Η Γενική Διεύθυνση για τη Διεύρυνση όμω ή για την ε, εκπαίδευση χρησιμοποιούν ε, διαφορετικά έντυπα ε, και μερικοί από αυτούς χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα καταχώρησης. Διαφορετικά διοικητικά έγγραφα επίση, επειδή δεν χρησιμοποιούν πάντα το ίδιο σύστημα καταχώρηση. Πρέπει λοιπόν κανεί να τυπώσει όλα τα έγγραφα αυτά και να τα υποβάλει μαζί με την αίτηση. Οι βέλτιστε πρακτικέ από τη δική μα πλευρά είναι οι εξή. Θέλουμε, είμαστε υπέρ μια ε, βάση δεδομένων ε, επιγραμματική, όπου να μπορούν να ε, σώζονται τα έγγραφα, όπω γίνεται και στι περιπτώσει των δωρεών. Θέλουμε αυτό να γίνεται στου διαγωνισμού, γιατί αν κοιτάξετε το πρόγραμμα για την τεχνική βοήθεια, τα διοικητικά μα έγγραφα, ανέρχονταν σε 600 σελίδε, οι οποίε έπρεπε να αντιγραφούν τρει φορέ Μιλάμε για πολύ χαρτί, λοιπόν, πολύ σπατάλη χαρτιού και θα ήταν πολύ πιο εύκολο απλά να μπορεί να ανεβάσει κανείς τα έγγραφα αυτά στη βάση δεδομένων. Είμαστε υπέρ αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μια διαδικασία σε δύο στάδια και για τις δωρεές και για, τις, ε, ε, και για τους διαγωνισμούς. Ε, δηλαδή μια φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προέκυση και κατόπιν την αίτηση. Μας αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία και θα θέλαμε να διατηρηθεί. Και το τελευταίο θέμα που είναι μια πολύ δική περίπτωση είναι ότι επειδή ε, ε, απαιτεί η συμμετοχή ε, τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε από πριν ποιο είναι ο ρόλο των μη κυβερνητικών αυτών οργανώσεων, διότι γενικά δεν συμμετέχουν σε τέτοιου είδου διαγωνισμού οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και είναι πολύ δύσκολο να του εξηγήσουμε τι θα απαιτηθεί από αυτού αργότερα κατά τη διάρκεια τη διαδικασία. Όσον αφορά την εφαρμογή ε, για το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας, ε, η σύμβαση υπεγράφει τον ε, Δεκέμβριο. Αυτή τη βδομάδα θα υποβάλουμε μια έκθεση και οι πρώτες δραστηριότητε θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2013. Αλλά ήδη βλέπουμε από τις εμπειρίες μας στην αρχική φάση τέσσερα πράγματα θα ήθελα να αναφέρω. Ε, είχαμε μια αρχική φάση δίμηνη ε, που συμπεριλαμβανόταν στους όρους αναφοράς ε, και αυτό το βλέπουμε συχνά στους όρους αναφοράς για διαγωνισμούς. Οι δύο μήνε είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όμω και ακόμα και αν προτείνει κανεί μακρύτερο χρονικό διάστημα, αυτό δεν λαμβάνεται πάντα υπόψη. Ο ρόλος του εταίρου και η αποζημίωση για τις εργασίες στις περιπτώσεις αυτές ε, οι εταίροι είναι ε, ε, όπως οι κλασικοί εταίροι σε έναν όμιλο, αλλά από την άλλη απαιτείται να εργαστούν ως help desk, στα, γραφεία βοήθειας δηλαδή, στις χώρες τους. Όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ συχνά η διαδικασία αυτή κρατάει πολύ χρόνο, κατανοητό, αλλά δεδομένου του όγκου των αιτήσεων, αλλά ε, μερικές φορές είναι δύσκολο να πληρώσει κανείς εγκαίρως τους ε, εμπειρογνώμονες και να μπορέσει να ε, εκτελέσει τις δαπάνες. Και επίσης η, καταγραφή, η καταχώρηση των ε, προγραμμάτων ε, αποτελεί κάποια προκαλεί κάποια προβλήματα, διότι εμείς συνεργαζόμαστε με την ε, κοινωνία των πολιτών, ε, με οργανώσεις τη κοινωνίας των πολιτών, ε, που μερικές φορές δημιουργεί δυσκολίες όσον αφορά τις τράπεζες. Όσον αφορά τα προγράμματα ε, που έχουν να κάνουν με χορηγίε. Ε, έχουμε δύο που συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα για τον Κάφκασο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. Θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή του χρονοδιαγράμματο ε, στην περίπτωση του Καυκάσου λόγω τη διαμάχη Αζερβαϊτζάν-Αρμενία και στη Λευκορωσία λόγω τη γενική κατάσταση στη χώρα. Δεν πετύχαμε τα ίδια αποτελέσματα στο Αζερβαϊτζάν όπω και σε άλλε χώρε λόγω στην παρεμπόδιση κάποιων δραστηριοτήτων από το Υπουργείο Εκπαίδευση. Αλλά αυτό που μα βοηθάει σε αυτέ τι δύο περιπτώσει είναι ότι έχουμε πολύ, καλή, πολύ καλές επαφές με τις ε, αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έχουν βοηθήσει να λύσουμε προβλήματα. Όσον αφορά τα προβλήματα κατά την ε, εφαρμογή για το πρόγραμμα του Καυκάσου. Έχουμε το πρόβλημα Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας με τον Αγκόρνο Καραμπάχ και την ε, πολιτική κατάσταση του Αζερβαϊτζάν, διότι υπήρχαν φόβοι όσον αφορά τις συνέπειες της Αραβικής Άνοιξης και ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή νέων στα προγράμματά μας. Ε, και όσον αφορά το πρόγραμμα της Λευκορωσία. γενικά είναι χώρα με μεγάλες δυσκολίες και είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να ε, πληρεί κανεί τους όρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λόγω των συνθήκων. Είναι πολύ δύσκολο να λάβουμε αποδείξει επίσημε για όλες τις δραστηριότητε μας. Είναι χώρα που λειτουργεί με μετρητά, είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθούν χρήματα σε λογαριασμού. είναι δύσκολο να στείλουμε έγγραφα. Ε, πρέπει να ε, δημιουργηθούν πολλά μέτρα ασφαλείας και δεν έχει κανείς ε, οικονομική επισκόπηση του συνόλου του προγράμματος. Υπάρχει κατακαιρματισμός των λογαριασμών διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να γνωρίζουν όλοι την ακριβή οικονομική κατάσταση του συνόλου του προγράμματος. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο που να, τα γνωρίζει, όλα. Και για τα δύο προγράμματα όμως έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τις αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βέλτιστες πρακτικές που διαπιστώσαμε λοιπόν ε, ήταν ε, ότι όταν η διαχείριση ε, γίνεται από τις τοπικές αντιπροσωπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό λειτουργεί καλύτερα επειδή γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση επιτόπου. Βέβαια όλα εξαρτώνται από την προσωπική συμμετοχή των διαφόρων εμπλεκομένων αλλά αυτή είναι η εντύπωσή μας πολύ καλή πρακτική είναι και η ε, ευελιξία ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες, ε, διότι δεν χρειάζεται προηγούμενη έγκριση ε, κάθε δαπάνης από πριν. Για του ε, διαγωνισμού. Ε, χρειάζεται κάτι τέτοιο, το οποίο απαιτεί ε, σημαντική διοικητική προσπάθεια και πολύ καλή πρακτική. Είναι ο τρόπο που το Υπουργικό Συμβούλιο των Βορείων Χωνών παρέχει βοήθεια προς την Λευκορωσία. Πρόκειται για διακυβερνητική οργάνωση με βάση το Βίλνιους. Να συνοψίσω όσον αφορά τη χρηματοδότηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλου δωρητέ δεν είναι απαραίτητα επίκριση. Για, πολλού, για πολλές περιπτώσεις καταλαβαίνουμε τους λόγους, ε, αλλά μερικές φορές ε, δυσκολεύουμε τη ζωή για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, υπάρχει ε, λοιπόν, ε, σημαντικό άρθρος λόγω ε, των ε, απαιτήσεων που αυξάνονται ε, και υπάρχει ο κίνδυνος να απορριφθεί η αίτηση επειδή δεν ήταν τα καλή. Ε, επίσης, απαιτούνται συνέχεια όλο και περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων προς αντιπροσωπείες και το έντυπο για τον προϋπολογισμό δεν ε, καλύπτει απαραίτητα ε, τις ανάγκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι ο δικός μας προϋπολογισμός βασίζεται στις δραστηριότητες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί προϋπολογισμό ανά τύπο δαπάνης υπάρχει αυξημένος ανταγωνισμός ε, με την ίδια διαθεσιμότητα ε, πόρων, ε, το οποίο φυσικά δυσκολεύει την κατάσταση. Υπάρχει το ποσοστό διοικητικών ταπανών, 7% στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρκετά χαμηλό ποσοστό αυτό. Ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει προσαρμοστεί το ποσοστό αυτό. είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε το, ε, την συναλλαγματική ισοτιμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τη αγορά. Ε, να σα δώσουμε ένα παράδειγμα. Ολοκληρώνουμε ένα πρόγραμμα στη Μοζαμβίκη, ε, σχετικά μικρό πρόγραμμα, αλλά μετά από δύο χρόνια έχουμε απώλειες 9.000 ευρώ λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ε, και αυτό δεν μπορεί να το επιστρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του δημοσιονομικού κανονισμού. Υπάρχουν πολλές απαιτήσει όσον αφορά ε, την ε, λογιστική που δυσκολεύει τη ζωή για τις, τοπικούς, για τις τοπικές οργανώσεις και γενικά δεν έχουμε προγράμματα μακράς διαρκείας. Τρία με πέντε χρόνια συνήθως είναι το μέγιστο και δεν υπάρχει πολλή δυνατότητα για θεσμική υποστήριξη Και αν συγκρίνω την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με την γερμανική χρηματοδότηση, ε, ε, η ε, ανάθεση της σύμβασης είναι σχεδόν εξίσου δύσκολη, αλλά υπάρχουν λιγότερα εμπόδια. Είναι πιο ε, απλό το έντυπο, είναι πιο εύκολος ο προϋπολογισμός, ε, μπορεί να προσαρμοστεί από τον ε, Τούντα και είναι πιο εύκολο να καταλάβει κανείς ποια προγράμματα μπορούν να είναι επιλέξιμα, διότι φαίνεται τι προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί στο, μέλλον, στο παρελθόν και πού θέλουμε να κινηθούν στο μέλλον. Οι διοικητικές δαπάνες ανέρχονται σε υψηλότερο ποσοστό, 14% αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και ε, λαμβάνουμε και επιστροφή του ΦΠΑ. Και επίση ε, σημαντικό είναι ότι μπορεί να γίνει ε, θεσμική χρηματοδότηση, δεν χρηματοδοτούνται δηλαδή μόνο οι δραστηριότητε. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε και ευχαριστώ που κρατήσατε και τον χρόνο σα σχεδόν επανήλθαμε στο χρονοδιάγραμμα που έπρεπε να έχουμε τηρήσει. Και τώρα ο τελευταίος μας ομιλητής που είναι ο Ρίτσαρτ Μπέλς, επικεφαλής ε, του τμήματος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την ε, Ανατολική Εταιρική Σχέση. Έχεις το λόγο, Ρίτσαρτ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που έχω να μιλήσω στην Επιτροπή σας σήμερα. Καταλαβαίνουμε το απόλυτα το ενδιαφέρον της Επιτροπής να έχει μια γενική εικόνα για τη χρηματοδότηση για την ανατολική εταιρική σχέση και με ευχαρίστηση θα συμπληρώσω τις παρατηρήσεις του Μάρκου Κορνάρο. Θα ξεκινήσω όμω με μια προειδοποίηση για την υγεία, όπως ίσως γνωρίζετε βασικά από τα ε, οικοδομήματα που στηρίζουν το μέλλον δεν έχουν ακόμα φτιαχτεί, δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο βασικά και εξακολουθούμε να είμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά για τα εξωτερικά δημοσιονομικά μέσα όπως αυτό εδώ για το μέλλον. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να κάνω με την αδειά σας σήμερα είναι στο πρώτο τμήμα της παρέμβασής μου να πλαισιώσω πολιτικά τη συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί, να μιλήσω δηλαδή για τα επιτεύγματα και τον τρόπο που θα προχωρήσουμε στην ε, διάσκεψη κορυφής του Βίλνιους αργότερα ε, φέτος και γενικότερα μετά με γενικότερους όρους φοβούμε θα μιλήσω για το μέλλον και το νομισιονομική λογική πίσω από αυτά τα σχέδια για το μέλλον. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας περιγράψω Τι καταφέραμε εδώ και τέσσερα χρόνια, από τότε δηλαδή που δημιουργήθηκε στην διάσκεψη κορυφής της Πράγας το 2009 η Ανατολική Εταιρική Σχέση. Η ιδέα ήταν η σχέση ανάμεσα στην Ένωση και στους ανατολικούς της εταίρους να έρθει σε ένα άλλο επίπεδο μέσω της εμβάθυνσης ε, της ε, πολιτικής συνεργασίας αλλά και μέσω της δημιουργίας ενός πολυμερούς πλαισίου για συνεργασία και διάλογο. Διμερές επίπεδο καταρχήν. Ε, ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με πέντε από τους έξι εταίρους ώστε να θεσπίσουμε νέες συμβατικές σχέσεις με αυτές αυτές τις χώρες υπό τη μορφή των συμφωνιών σύνδεσης και με τέσσερις εξ αυτών των εταίρων αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, ολοκληρώθηκαν με συνομιλίες για βαθύτερες ε, ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Πρόκειται για τις ε, πιο εις βάθος συμφωνίες που έχει κάνει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση με ε, εταίρους ολόκληρο τον κόσμο. Η συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία ήταν θέμα στις 1η ε, Μαρτίου του 2012 και η σχετική συμφωνία με την Μολδόβα, την Γεωργία και την Αρμανία είναι κοντά στην ολοκλήρωσή τους αυτή τη στιγμή, ενώ οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης με το Αζερβαϊτζάν επίσης έχουν ξεκινήσει. Ένα δεύτερο στοιχείο πολιτικής σύνδεσης και οικονομικής ολοκλήρωσης είναι η ιδέα ενθάρρυνσης μεγαλύτερης κινητικότητας και επαφής μεταξύ των ανθρώπων εντός της ε, ανατολικής εταιρική σχέσης και εκεί έχουν ληφθεί μια ολόκληρη σειρά από μέτρα. Έχουμε διευκόλυνση βίζας και επανεισδοχής με την Μολδόβα, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Ε, Διευκόλυση επίσης, συμφωνία διευκόλυνσης ε, θεωρήσεων με την Αρμενία έχει υπογραφεί και έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Αζερβαϊτζάν. Η προσφορά για διαπραγμάτευση παρόμοιες, παρομοίων μάλλον διευκολύνσεων με τη Λευκορωσία έχουν ξεκινήσει από το 2012, αλλά προς λύπη μας αυτή η προσφορά δεν έχει γίνει δεκτή για την ώρα από τις αρχές του Μίνσκ. Επιπλέον, ε, εταιρικέ σχέσεις κινητικότητας με κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει με την Γεωργία, Μολδόβα και Αρμενία και ακόμη πιο σημαντικό, απελευθέρωση, μάλλον προγράμματα δράσης για την απελευθέρωση των θεωρήσεων έχουν ξεκινήσει με την Μολδόβα, τη Γεωργία και πιο πρόσφατα με την Γεωργία ε, για να προετοιμαστεί το έδαφος για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των θεωρήσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ιδρικής Όπως είπε και ο Μάρκος σήμερα το πρωί, αυτή η διμερής ατζέντα έχει συνοδευτεί από σημαντική οικονομική στήριξη. Για να σας τονίσω κάτι που δεν νομίζω πως αναφέρθηκε σήμερα το πρωί και που επίσης σχετίζεται με ένα σχόλιο προηγούμενο μιλητή, τα προγράμματα, τα συνολικά προγράμματα οικοδόμηση θεσμών είχαν σχεδιαστεί για να στηρίξουν τις χώρες εταίρου και τους διοικητικού του μηχανισμού στι διαπραγματεύσεις αυτών των κειμένων και την εφαρμογή των δεσμεύσεων, την υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτέ τι συμφωνίες. Και θα πρέπει να πω ότι σε σχέση με αυτά τα προγράμματα και ιδιαίτερα ε, υπήρξαν ε, θεατικοί και εκτεταμένοι διάλογοι ανάμεσα στους διαπραγματευτές μας επιτόπου και στις χώρες εταίρους. Οπότε πραγματικά έχω ένα αριθματολόγιο σε σχέση με ένα από τα σχόλια και την, που αφορούσε την ετοιμότητα των δικών μας αντιπροσωπιών να εμπλακούν σε σοβαρό διάλογο με τις χώρες εταίρους. Η δική μου εντύπωση δεν είναι αυτή πάντως. Τώρα, στο πολυμερές μέτωπο έχουμε την αρχιτεκτονική που χρειάζεται, έχουμε διασκέψεις κορυφής κάθε δύο χρόνια, επαφές των, συνδιασκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών κάθε χρόνο, έχουν επίσης θεσπιστεί ε, συνεδριάσεις των ανώτατων ε, υπαλλήλων και συνεργασία σε, πολλές, ε, σε πολλούς τομείς πολιτικής, ώστε να υπάρχει μόνιμος διάλογος ανάμεσα στους εταίρους με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλύτερων πρακτικών και όπως ήδη έχει αναφερθεί συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ένωσης που έχουν πρόσφατες εμπειρίες από την μετάβαση τα ίδια σε σχέση με την προσέγγιση δηλαδή των προδιαγραφών της Ένωσης. Πιο τελευταία φτιάξαμε και την, τον άτυπο, τους άτυπους διαλόγους με τους ανατολικούς εταίρους ανάμεσα δηλαδή στους έξι υπουργούς εξωτερικών των χωρών εταίρων και πιο πρόσφατα στη Γεωργία. Αυτό το επεκτείναμε και σε συζητήσεις για συγκεκριμένους τομείς, για τις μεταφορές συζητήσαμε το Φεβρουάριο. Αυτές οι πολυμερείς δραστηριότητες τονίζονται από διάφορες ε, βασικές πρωτοβουλίες ε, που τις περιέγραψε σήμερα ε, το πρωί ο Μάρκος, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Ένα από τα κλειδιά της εταιρικής σχέσης αυτής ήταν η προσπάθεια να φτάσουμε στις κυβερνήσεις και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μεταρρυθμίσεων που απαιτούν την εμπλοκή όχι μόνο των κυβερνήσεων και των διοικητικών δομών, αλλά και της κοινωνίας πλατύτερα. Ε, είμαστε λοιπόν ευχαριστημένοι που οι οργανώσεις ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών στην Ένωση αλλά και στις χώρες εταίρους έχουν φτιάξει τα αντίστοιχα φόρουμ που τώρα έχουν επεκταθεί και σε εθνικό επίπεδο μέσω της δημιουργίας εθνικών βάσεων για την κοινωνία των πολιτών και το διάλογο που νομίζω ε, βοηθούν να μετρήσουμε την εμπλοκή και την εφαρμογή των νέων συμφωνιών από τους εταίρους μας και είναι ένα κλειδί για να ενθαρρύνουμε τον ε, κοινωνικό διάλογο ανάμεσα στους ε, εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Εσείς ως ευρωβουλευτές έχετε πολύ σημαντικό ρόλο να παίξετε, πιστεύουμε, στην ε, Ανατολική Εταιρική Σχέση, γιατί είμαστε ευχαριστημένοι που η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest έχει πλέον θεσπιστεί και θα κάνει την επόμενη τη συνεδρίαση τον Μάιο φέτος και παρομοίως σε επίπεδο τοπικών αρχών η διάσκεψη Κόλυπ ε, στη διάσκεψη δηλαδή των εταίρων ανατολικής εταιρικής σχέσης έχει πλέον ε, εγκαθιδρυθεί. Όπως είπα, δύο χρόνια πέρασαν, ε, τέσσερα χρόνια συγγνώμη, πέρασαν από την Πράγα και εντός της Ένωσης έχουμε αρχίσει να προετοιμαζόμαστε για τη διάσκεψη κορυφής του Βίλνιους που προβλέπεται για τον Νοέμβριο. Έγινε σχετική συζήτηση στο Υπουργού Εξωτερικών φέτο, και ε, συμπεριλαμβάνεται το θέμα και στα πορίσματα του Συμβούλιο. Είναι μια καλή ευκαιρία ώστε να, θα τοποθετηθεί ένας ακόμα, ένα ακόμα ορόσημο θα μπορούσε να αποκλειθεί μάλιστα και η διάσκεψη κορυφή ε, τη απόδοση ε, των αποτελεσμάτων και αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από την ετοιμότητα των κρατών ε, αυτών να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις. Ελπίζουμε ότι μέχρι να έρθει η ώρα για το Βίλνιους θα έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Η Ουκρανία από την πλευρά της ξέρει τι χρειάζεται να κάνει για να μπορέσει η Ένωση να υπογράψει την Συμφωνία Σύνδεσης στο Βίλνιους. Αυτά όλα αναφέρονται στα συμπεράσματα του Υπουργείου Εξωτερικών υποθε... των... της διάσκεψης μάλλον των Υπουργών Εξωτερικών του Δεκεμβρίου και η συμφωνία σύνδεσης με τη Μολδόβα, τη Γεωργία και την Αρμενία θα ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι. Και επίσης στον τομέα της κινητικότητας θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δείξουμε καλή πρόοδο προς την απελευθέρωση των θεωρήσεων Είμαστε επίση πεπισμένοι πως θα έχουμε προχωρήσει και στην ε, διαπραγμάτευση των ε, ημερησίων διατάξεων σύνδεσης που θα είναι μια νέα γενεά σε σχέση με τα προγράμματα δράσης και θα έχουν σχεδιαστεί ώστε να προετοιμαστεί και να, εφαρμοστεί, να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν οι νέες συμφωνίες. Επίσης στο Βίλνιος περιμένουμε πρόοδο στον τομέα των μεταφορών όπου συνεχίζεται η δουλειά για να υπάρξει ένα ε, δίκτυο μεταφορών της ανατολικής εταιρικής σχέσης που θα συνδέει του χώρες εταίρους με το δίκτυο TEN-T της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά συζητήθηκαν και στη στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής της ε, Βαρσοβίας και μάλιστα οι Λιθωνοί προετοιμάζουν ένα, επίσης, ένα ακόμα φόρουμ επιχειρήσεων ώστε να συνδεθούν όλα αυτά με την ατζέντα της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό γιατί ελπίζουμε πως θα έχουμε ε, συμφωνίες βαθύτερων ε, εμπορικών συναλλαγών, ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών σύντομα. Έχει λοιπόν στρωθεί ο δρόμος για την ατζέντα του μέλλοντος. Έχει γίνει η πορεία πια αυτή είναι μία αναστρέψιμη για την οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση. Αυτή η διαδικασία για το μέλλον όπως ήδη τονίστηκε και το πρωί πιθανότατα θα διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις ε, χώρες εταίρους. Από τη μια πλευρά Θέλουμε να πάμε όσο γίνεται πιο, να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και να στηρίξουμε τις χώρες αυτές με ισχυρέ φιλοδοξίε, ενώ ταυτόχρονα η, ανατολική εταιρική σχέση θα πρέπει να παραμένει πλαίσιο και για εκείνους που ακολουθούν πιο αργό μονοπάτι μεταρρύθμισης που δεν έχουν βλέψεις για να προσχωρήσουν στην Ένωση. Πάντως, σε περαιτέρω εξελίξεις ε, στις σχέσεις της Ένωσης θα απαιτήσουν περισσότερη δράση σε τρεις σημαντικούς τομείς, ε, μια πλήρως, ένα πλήρως λειτουργών δικαστικό σώμα, αποτελεσματική δημόσια και πρόοδος προς την εκρίζωση του, της διαφθοράς. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό όσον αφορά την χρηματοδότηση για το μέλλον. Καταρχήν να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες της Κομισιόν σε κάθε δραστηριότητα προγραμματισμού. Δουλεύουμε σε στρατηγικό επίπεδο όσον αφορά τα πολιετή έγγραφα στρατηγικής και τα ενδεικτικά προγράμματα. Με χαρά επίσης μπορώ να σας πω ότι αυτή η διαδικασία συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Επιτροπής όπως ισχύει για το Ευρωπαϊκό Μέσο Γεννίασης είναι εξαιρετικά παραγωγικό. Και τώρα να πω δύο λόγια για την λογική την πολιτική που διέπει το Ευρωπαϊκό Μέσο Γετνίαση Η βάση για τη δουλειά μας, όπως είπαμε και το πρωί, είναι η το, το ανακοινωθέν Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γετνίασης του 2011 που εκθέτει την αναθεωρημένη πολιτική ε, γετνίασης. Υπάρχουν δύο σημαντικά και έννοιες που προκύπτουν από αυτό το ανακοινωθέν αυτήν την ανακοίνωση όσον αφορά τις δημοσιονομικές δραστηριότητε για το μέλλον. Το πρώτο είναι αυτή η έννοια ότι θα πρέπει να ε, στηριχτούν οι εταίροι που, το, ε, που δημοκρατία όπως ε, ονομάστηκε τότε αυτή η διαδικασία και να έχουμε και μια προσέγγιση more for more. Η ανακοίνωση υποδεικνύει ότι θέλουμε να απλοποιήσουμε την πολιτική και το πρόγραμμα πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ότι χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό, μάλλον μια νέα γενεά σύνδεσης, συμφωνιών σύνδεσης, δηλαδή πολιτικά μηνύματα για νέες συμφωνίες συνδυασμένα με ένα ενιαίο πλαίσιο στήριξης που συνδυάζει τα όσα γίνονταν στο παρελθόν μέσω ενός εγγράφου στρατηγικής για τη χώρα και ενός ε, πολιετούς, ε, ενδεικτικού πολιετούς προγράμματος. Όλα αυτά λοιπόν συμπεριλαμβάνονται στο μέσο για την ευρωπαϊκή πολιτική κοινωνία που είναι επιτάπητος. Όποιε και αν είναι οι συγκεκριμένε προτεραιότητε λοιπόν, που θα έχουμε για κάθε μια από αυτέ τι χώρε εταίρου στο μέλλον, υπάρχουν τρει βασικοί τομεί όπου περικλείεται η συνεργασία με τους εταίρους μας. Καταρχήν θέλουμε να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τη διαδικασία πολιτικής σύνδεσης και οικονομικής ολοκλήρωσης. Δεύτερον, θέλουμε να ε, αυξήσουμε τις προσωπικές επαφές και να ε, έρθουμε σε επαφή ευρύτερα με την κοινωνία και να στηρίξουμε τομείς κλειδιά για την οικονομική ανάπτυξη. Οι μικρομεσαίες είναι μία προφαν... ένας προφανής τομής, τομέας, ε, η γεωργία άλλος και επιπλέον τομείς κλειδιά όπου η διασύνδεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους θα είναι πολύ σημαντική. Οι μεταφορές και η ενέργεια είναι φυσικά ε, τομείς κλειδιά. Όπως είπα, Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τα νέα μέσα, οπότε δεν μπορώ να μπω σε πολλές λεπτομέρειες για να σας παρουσιάσω αυτά τα σχέδια που έχουμε για το μέλλον, αλλά να πω ένα-δυο πράγματα ωστόσο. Καταρχήν δεν πιστεύω πως προβλέπεται αλλαγή στη δομή των προγραμμάτων σε σχέση με τα ισχύοντα, με την έννοια ότι θα έχουμε διμερεί προγράμματα με κάθε μια από τις χώρες εταίρους, θα έχουμε ένα φάσμα εθνικών προγραμμάτων και θα έχουμε και διασυνοριακή συνεργασία. Η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο μέσο πιθανότατα θα είναι σε διμερές επίπεδο. Ήδη αναφέραμε τη σημασία μεγαλύτερης ε, στόχευσης της βοήθειάς μας. Αυτό θα είναι ένας στόχος που θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε στα πλαίσια ενιαίας στήριξης που θα είναι προγραμματικά έγγραφα για μεμονωμένες χώρες εταίρους. Έχουμε ήδη ξεκινήσει αρχικές επαφές μέσω των αντιπροσωπιών μας με τις χώρες εταίρους για να εντοπίσουμε ναι, κάποιους συγκεκριμένους τομείς που μπορούμε να στηρίξουμε στο μέλλον. Και σε διμερές επίπεδο πιστεύω πως η έννοια μιας προσέγγισης με βάση κίνητρα θα είναι πιο ορατή. Οι συζητήσεις για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό συνεχίζονται. Α, θα σας πω ότι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας θα, θα, θα ε, εισαχθεί ένα στοιχείο κινήτρου σε σχέση με τις αρχικές ε, τα αρχικά ποσά αναχώρα θα, θέλουμε να θα θελήσουμε να εξασφαλίσουμε πως αυτά τα ποσά προσωπεύουν, αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση των χωρών να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και το επίπεδο φιλοδοξίας ε, που έχουν για τις σχέσεις τους με την Ένωση. Μέσω, κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περίοδου θα ε, προβλέψουμε και τη δυνατότητα ευελιξίας όσον αφορά τα κονδύλια ανά χώρα ώστε να προσαρμόζονται τα ποσά ανάλογα με την πρόοδο. Και όπως ανέφερε ο Μάρκους, Ήδη έχουμε υπό την ισχύουσα συμφωνία κάποια προγράμματα με βάση κίνητρα όπως τα, που τα λέμε ΙΠΕΚ, και που θα εξακολουθήσουν να παρέχουν κίνητρα για τις χώρες που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά βέβαια θα παρακολουθούνται μέσω της αιτήσιας έκθεσης πρόοδου που προετοιμάζεται για κάθε μία χώρα όπου υπάρχει ατζέντα σύνδεσης ή πρόγραμμα ε, εταιρικής σχέσης. Για να καθορίσουμε πώς θα κρίνουμε κάθε φορά τη χώρα, πώς έχει αποδώσει και αυτό θα παίξει ρόλο κλειδί για την απόφαση για την ε, κατανομή χρημάτων. Αυτά για το διμερές επίπεδο. Στο πολυμερές επίπεδο προβλέπουμε μια παρόμοια ρύθμιση με αυτή που ισχύει σήμερα, δηλαδή ένα πρόγραμμα περιφερειακό μέσα στο πλαίσιο της ε, πολιτικής γετνίασης. Ο Μάρκος ανέφερε την διευκόλυνση ε, γετνίασης για τις επενδύσεις, ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες. Επειδή θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιφερειακό προς Ανατολάς που θα προσπαθήσει να κάνει πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν μέσω των διμερών προγραμμάτων και των σχετικών εγγράφων. Και μία από τις πτυχές κλειδιά εδώ είναι να στηριχθούν η, να στηριχθεί η πολυμερής διαδικασία της ανατολικής συνεργασίας Επίσης να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή την έννοια των πρωτοβουλειών ε, ναυαρχίδων, των βασικών δηλαδή ε, πρωτοβουλειών. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή ποιες θα είναι οι επόμενες, να δούμε ποιες θα είναι οι, δυνατότητες για το μέλλον. Είναι ένας τομέας όπου συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη ώστε να ενσωματώσουμε ενδεχομένω ιδέες τους. Τέλος, διασυνοριακή συνεργασία και σχετικά προγράμματα που θα συνεχιστούν ως ένας ακόμα τρόπος για στήριξη της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Η σημασία της συνεργασίας με τα άλλα μέσα ήδη αναφέρθηκε σήμερα το πρωί και ενώ το μέσο Ευρωπαϊκής Γετνίασης θα είναι το βασικό μέσο για τη στήριξη της ανατολικής εταιρικής ε, σχέσης, εμείς στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μαζί με τους συναδέλφους της Υπηρεσίας της Κομισιόν θα θέλαμε ο προγραμματισμός μας να λαμβάνει υπόψη τα άλλα μέσα τα οποία ισχύουν για το μέλλον. Τόσο τα, εσωτερικά και τα, όσο και τα εσωτερικά. Στα εξωτερικά έχουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το μέσο για τη σταθερότητα και το μέσο για την συνεργασία και την πυρηνική ασφάλεια όπου όλα αυτά θα συνεχίσουν να παίζουν ρόλο για την ε, ανατολική εταιρική σχέση καθώς και κάποια θεματικά προγράμματα υπό το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα μέσα εξωτερικής συνεργασίας, ε, αλλά και εσωτερικά μέσα θα είναι σημαντικά για το μέλλον της ανατολικής εταιρικής σχέσης επίσης, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την εξωτερική συνεργασία όπως ε, το Connecting Europe, το Creative Europe και το Horizon 2020. Τώρα, εκτός του πλαισίου των ευρωπαϊκών μέσων, είναι σαφές ότι και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία θα είναι ένα μέσο για τη στήριξη των ευρωπαϊκών στόχων στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία μετάβασης, μεταρρύθμισης παίρνει χρόνο και αυτό το μέσο είναι σχετικά νέο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Ελπίζουμε ότι μέχρι το Βίλνιος θα έχουμε μια νέα γενεά συμφωνιών με τις χώρες εταίρους και θα έχουμε ένα σαφέστερο πλαίσιο για αυτή την μεταρρύθμιση. Και η οικονομική μας στήριξη για την Ανατολική Εταιρική Σχέση για το μέλλον θα σχεδιαστεί ώστε αυτές οι διαδικασίες μετάβασης να προχωρήσουν. Εμείς θα θέλαμε να σημειωθεί συμφωνία σύντομα στο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη δουλειά μας, όπως θα θέλαμε και να βρεθεί συμφωνία για τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης, ώστε σύντομα να προχωρήσουμε με τον προγραμματισμό από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η νέα δημοσιονομική περίοδος το 2014. Σας ευχαριστώ. Uh, εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Φυσικά όλοι επιθυμούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθεώρησης ε, όσο δυνατόν πιο σύντομα. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές μας που τήρησαν και το χρόνο τους. Δύο έχουν ζητήσει τον λόγο. Οποιοςδήποτε άλλος παρακαλώ να μας ενημερώσει. Πρώτος ο Σάιρους Βόλσκι. Ευχαριστώ. Λέει ο Βόλσκι. Η ερώτησή μου είναι, έχοντας ακούσει όσα υπόθηκαν, γιατί κάνουμε τόσο πολλά με τόσο πενιχρά αποτελέσματα. Επειδή είμαι τώρα και στο Euronest και έχω λάβει και εγώ ε, βοήθεια στο παρελθόν, με τρομάζει το πόσο εφησυχάζουν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η αντίθεση με αυτά που λένε αυτοί που είναι επιτόπου. Στην πράξη φαίνεται τι έχουμε κάνει και κινδυνεύει να καταρρεύσει η σχέση μας αυτή και σε πολλές χώρες Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία έχουμε ε, υποχωρήσεις στην πρόοδο της δημοκρατίας αφού έχουμε όλα αυτά τα θαυμάσια όργανα. Γιατί αποτυχάνουν οι πολιτικοί μας στόχοι. Τι προκύπτει από αυτά που ακούμε, ε, ε, βοήθεια για την ανάπτυξη, για την προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο, αλλά υπάρχει πολύ έλλειψη αποτελεσματικότητας στις δράσεις μας. Ως ε, μέλος της ΑΦΕΤ, η άποψη του Κοινοβουλίου για το κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι στην πολιτική ανατολική γειτονία είναι τελώς διαφορετική από αυτήν την ε, απόλυτη ικανοποίηση που διαπιστώνουμε από τις διάφορες υπηρεσίε, ιδίως την ΤΕΒΚΟ. Η βοήθεια αυτή είναι υπερβολικά κατακαιρματισμένη. Είναι μια βοήθεια τούτη φρούτη που δεν μπορεί να επιτύχει. Δίδονται μικρέ χρηματοδοτήσει ε, κατατέμνονται ακόμη περισσότερο για μια πληθώρα προγραμμάτων, προγραμμάτων τα οποία κανείς δεν μπορεί να παρακολουθήσει και να καταλάβει. Η Ένωση δεν έχει επαρκή ποσά για να καλύψει όλα αυτά που θα ήθελε να κάνει. Αναπτυξιακή, βοήθεια εξυγχρονισμού, προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε και, αυτούς, αυ, και τους τρεις αυτούς στόχους. Μπορούμε να δώσουμε κάποια βοήθεια για προσαρμογή στην Ένωση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις. Λυπάμαι πολύ που οι υπηρεσίες δεν εξάγουν διδάγματα από την αποτυχία των χρηματοδοτήσεων που δόθηκαν στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης πριν από 10 περίπου χρόνια. Ακούγοντας αυτά που υπόθηκαν σήμερα, έχω την αίσθηση ότι τα έχω ξανακούσει όλα αυτά. Τα ίδια λάθη, τα ίδια παράπονα, τα ίδια δόγματα που αντιμετωπίσαμε όταν ήμασταν υπό ένταξη χώρες στη δεκαετία του 90. Είναι κρίμα. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά. Οι πόροι αυτοί δεν είναι δυνατόν να μετατρέψουν όλη αυτή την περιοχή και να προκαλέσουν τεράστια αλλαγή τύπου Big Bang. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είπε «Ε, χρειαζόμαστε χρόνο. Αλλά εντωμεταξύ η Ρωσία ανακαταλαμβάνει τα μετασοβιετικά κράτη. Τα προγράμματα αυτά δημιουργούν αυταπάτες ότι θα αλλάξει η κατάσταση στην Ανατολή. Αλλά η ομή πραγματικότητα είναι ότι χάνουμε τους ανατολικούς γειτονές μας. Αυτή η προσέγγιση περισσότερα για περισσότερα ότι όποιος ε, δηλαδή πάει καλά πρέπει να πάρει επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Μα δεν υπάρχουν επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Και το θεσμικό πλαίσιο με ανησυχεί. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο δεν λειτουργούν σωστά οι υπηρεσίες της Κομισιόν και της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και δεν ανταποκρίνονται στα όσα έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο όταν δημιουργήθηκε αυτή η πολιτική και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και υπενθυμίζω ότι όταν δημιουργήσαμε το ΦΑΡ στη δεκαετία του 90 η βοήθεια πήγε στην ΡΕΛΕΞ και όσοι θυμούνται θυμούνται ότι μόνο μία γενική διεύθυνση ε, χορηγούσε αυτή τη βοήθεια και τα νούμερα που αναφέρθηκαν καταδεικνύουν ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Θα είχα και ερωτήσει για το πώς ε, αποφασίζονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις, αλλά εγώ ως συντονιστής της βοήθειας ε, της Ένωσης και του G24 στο παρελθόν ξέρω ότι τα ποσά αυτά προσθέτουν αχλάδια με μήλα και στην ουσία είναι αποτέλεσμα δημιουργικής λογιστικής. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Τατζίνσκα. Η βοήθεια πρέπει να βασίζεται στην ε, ζήτηση. Η μορφή της βοήθειας πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτούς που θέλουν να τη χορηγήσουν. Και πολύ συχνά ένα μεγάλο τμήμα αυτής της βοήθειας δεν μπορούμε κατόπιν να δούμε πού πήγε. Επειδή εμείς λαμβάναμε τότε, στη δεκαετία του 90, ε, βοήθεια, την καλούσαμε τότε βοήθεια μπούμεραγκ. Δηλαδή, ερχόταν σε εμά και ξαναγύρναγε στο χωρικό. Με τόσο λίγα χρήματα, ούτε αναπτυξιακή βοήθεια, ούτε επενδύσεις. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε ψάρια, μπορούμε να τους δώσουμε μόνο καλάμι για να ψαρέψουν και να μην έχουμε συγκαταβατική άποψη έναντι των ε, παραληπτών. Χρειάζεται διάλογος πριν σχεδιαστεί η βοήθεια. Αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Τατσίνσκα. Συνολικά θεωρώ ότι και οι στόχοι και οι μέθοδοι πρέπει να αναθεωρηθούν ριζικά μετά από διάλογο με τους παραλήπτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Γκέραν Φάρμ. Να μιλήσει και αυτός και μετά θα ζητήσουμε οι δύο οργανώσεις ε, ε, προς τις οποίες απευθύνθηκε ο Σάιρους θα πρέπει να απαντήσουν. Ευχαριστώ. Ήμουν εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών για μια γνωμοδότηση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και είμαι και συμπροέδρος ε, της Οικονομικής Επιτροπής του Euronest. Συζητήσαμε αναλυτικά το πώς λειτουργεί η συνεργασία σε αυτήν την Οικονομική Επιτροπή του Euronest. Έχουμε ήδη εγκρίνει μια έκθεση για σφαιρικές και βαθιές οικονομικές συμφωνίες. Συζητάμε και μια έκθεση για τις υποδομές μεταφορών, ε, πληροφορική, τεχνολογία κτλ. Όλα τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά δεν είμαι τόσο ριζικά επικριτικός όπως ο κύριος Βόλσκι, αλλά έχω και ερωτήσει και σχόλια. Πρώτον, η προσέγγιση περισσότερο για περισσότερο. Όλοι συμφωνούμε ότι με βάση και την πείρα μας με την Αραβική Άνοιξη, όπου προφανώς αποτύχαμε στην ενίσχυση της δημοκρατίας, αποτύχαμε στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξαναδούμε τι σημαίνει αυτή η θέση προϋποθέσεων. Ο κύριος Βόλσκι λέει πώς μπορούμε να, λούμε, να πούμε περισσότερο για περισσότερο όταν δεν υπάρχουν περισσότερα να δώσουμε. Ίσως ήταν καλύτερα να πούμε λιγότερο για λιγότερο. Δηλαδή, εάν κάποια ενίσχυση που δεν αξιοποιείται ορθώς, πρέπει να ε, καταργηθεί. Δεύτερον, οι σαν αναχώρα αλλά και χορηγήσεις ε, Ανατολή και Νότος. Η γνώμη της Επιτροπής Προπολογισμών τονίζει την ανάγκη μακροπρόθεσμης στρατηγικής χορηγήσεων. Αλλά χρειαζόμαστε βεβαίως και ευελιξία, διότι υπάρχει μια πολύ ειδική κατάσταση, για παράδειγμα στη Βόρεια Αφρική που χρειάζεται συμπληρωματική βοήθεια, τότε θα πρέπει να μπορεί να δοθεί. Ποια όμως είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ μακροπρόθεσμου, προβλέψιμου προγραμματισμού και ευελιξίας. Δεν είναι εύκολη η επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Τρίτον, ε, επενδύσεις και ενισχύσεις για ενίσχυση της δημοκρατίας. Οι επενδύσεις είναι βέβαια πάντα πολύ ελκυστικές ως τμήμα της αναπτυξιακής βοήθειας. Δίνουμε πολλά λεφτά και είναι ιδιαίτερα ορατά τα αποτελέσματα. Αν χτίσουμε ένα δρόμο, ένα αεροδρόμιο, μια μονάδα παραγωγής ενέργειας. Αλλά πρέπει να υπάρχει και άλλου είδου στήριξη, τεχνική βοήθεια, προώθηση της συμμετοχής ε, στα ενωσιακά προγράμματα, συμμετοχή στην εργασία των υπηρεσιών της Ένωσης και των οργανισμών ανάπτυξη δεξιοτήτων και άλλες μορφές κατάρτισης και αυτά είναι επενδύσεις, ζωτικές επενδύσεις. Και επίσης, συγκεντρωτισμός ή αποκεντροποίηση, γιατί σε πολλές μετακομμουνιστικές χώρες υπάρχουν πολύ συγκεντρωτικές δομές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, οργανώσεων κοινότητα των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πολύ σημαντικό αυτό. Συνεργαζόμαστε βεβαίω με τι κυβερνήσει. Αλλά οι κυβερνήσει κυρίω ενδιαφέρονται για συγκεντρωτικού τύπου ανάπτυξη. Δεν βοηθάνε τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν διδημοποίηση θα πρέπει να έχουν και αυτό το στόχο. Τέλος, κατακαιρματισμό πληθώρα προγραμμάτων. Βεβαίω ε, πέρυσι το συζητήσαμε όταν συζητούσαμε τη νέα χρηματοδότηση για τη δημοκρατία, το νέο ταμείο για τη δημοκρατία. Ήδη όμως είχαμε ένα μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς λοιπόν να αποφύγουμε επικάλυψη μεταξύ αυτών των δύο. Ένα μόνο παράδειγμα. Σε πολλούς τομείς πρέπει να ξαναδούμε τους κινδύνους επικαλύψεων. Ιδιαίτερα, όπως είπαμε στην ονομοδότησή μας, να δούμε και το συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Γιατί δεν υπάρχει μόνο η Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν και διμερεί προγράμματα ενίσχυσης. Άρα χρειάζεται συντονισμός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Συντόνια. Για μένα αυτή η ακρόαση δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις, αλλά ίσως και αυτό είναι θετικό. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω στα αρχικά ερωτήματα που έθεσα και στην Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κατά την προετοιμασία αυτής της ακρόασης, διότι κάποιες από τις παρατηρήσεις των δύο συναδέρφων μου μπορεί να μην είναι ερωτήσεις ε, προς τους παρόντες, ε, μπορεί να έχουν να κάνουν ε, με το πολιτικό θεματολόγιο και θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε τους παρόντες τι μπορούν να μας απαντήσουν. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που συνδέονται Ε, με την Κομισιόν. Καταρχήν προς τον κύριο Κορνάρο. Εκτιμώ τις προσπάθειές σας που ήρθατε εδώ και μας εξηγήσατε διάφορα πράγματα. Από πλευρά του προϋπολογισμού όμως δεν είμαι ικανοποιημένη και προφανώς ε, θα γνωρίζετε γιατί. Διότι υπάρχει ε, αρκετή σύγχυση ανάμεσα στις πιστώσει και στις πληρωμές. Είναι εξαιρετικό το ότι δεσμεύετε τόσα χρήματα. Πώ όμω μπορείτε να πληρώσετε. Χωρί μικρόφωνο. Προ τον κύριο Κορνάρο, για μένα είναι ενδιαφέρον από πλευρά του προπολογισμού να γνωρίζω πόσα χρήματα έχουν πληρωθεί, διότι τι πιστώσει υποχρεώσεων μπορώ να τι βρω στην ιστοσελίδα ε, σα. Ε, μπορώ να το βρω αυτό και χωρί βοήθεια. Αλλά όσον αφορά τι πληρωμέ, ε, υπάρχει κάποιο μυστήριο, διότι στην παρουσίασή σα είπατε ότι υπάρχουν πιστώσεις ε, υποχρεώσεων 2,8 δις. Εγώ θα ήθελα να ξέρω πόσα έχετε δαπανίσει αυτά τα χρόνια. Εάν δεν μπορείτε να δώσετε τις πληροφορίες τώρα, που από μόνο του πιστεύω ότι αποτελεί πρόβλημα, θα πρέπει να μας ε, υποβάλλετε γραπτό στην απάντηση ότι ε, τα μέλη της Επιτροπής μας πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο πόσα χρήματα υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πόσα δαπάνησε. όσον αφορά το διάστημα 2009-2012. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχετε και τα στοιχεία του 2012, αν όχι πλήρη, τουλάχιστον ε, εν μέρη πλήρη. Επίσης, όσον αφορά την αρχή more for more, περισσότερα για περισσότερα, ε, ε, θα ήθελα να, να μου το αναπτύξετε αυτό, θα ήταν ενδιαφέρον να το γνωρίζουμε. Και Ανησυχώ πολύ περισσότερο όσον αφορά την παρουσίαση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Για μένα δεν αποτελεί επιχείρημα το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει. Το γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ που μας το είπατε. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά θα πρέπει ήδη να έχετε προγραμματίσει τα επόμενα χρόνια. Συγγνώμη, αλλά σε τέσσερα χρόνια πρέπει να υποβάλλετε το σχέδιο προπολογισμού για το 2014. Νομίζω ότι μα αξίζει να λάβουμε πληροφορίε σχετικά με το προ τα που κινείστε. Επιμένω λοιπόν και σε αυτό να απαντήσετε γραπτό μετά τη σημερινή συνεδρίαση. Η σημερινή συνεδρίαση είναι πολύτιμη από μόνη τη, ελπίζω όμως ε, να ε, οδηγήσει και σε συλλογή πληροφοριών ε, για τους ευρωβουλευτές αλλά και για άλλους ενδιαφερομένους. Και είναι απαραίτητο να υπάρχει μια επισκόπηση του προγραμματισμού. Ελπίζω να πετύχουν οι διαπραγματεύσεις. Θα δούμε ποια θα είναι ε, τα αποτελέσματα, αλλά ήδη γνωρίζουμε τα νούμερα. Δεν πιστεύω ότι δεν έχετε κάνει τίποτα από τον Φεβρουάριο και μετά που συναντήθηκαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και συζήτησαν το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν έχετε προσαρμόσει τα αρχικά σα νούμερα και ότι δεν εργάζεστε πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό απλά δεν το πιστεύω. Θα έπρεπε λοιπόν ήδη να έχουμε λάβει τι πληροφορίε αυτέ και δεν τι έχουμε λάβει και ε, αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα λύπηρο. Και βέβαια δεν μπορώ να θέσω συγκεκριμένε ερωτήσει, διότι δεν είπατε κι εσεί τίποτα συγκεκριμένο σχετικά με το 2014 ε, με 2020. Ωστόσο, θα με ενδιέφερε να μάθω την άποψη των ομιλητών ε, σχετικά με το νέο Ταμείο για τη Δημοκρατία. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις παρατηρήσεις σας, διότι πρόκειται για νέο μέσο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Συντόνια. θα δώσω το λόγο μετά στους ε, ομιλητές για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ω μέλο της επιτροπή Πολιτισμού και εκπαίδευση θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Σε, πολλές, σε πολλά από τα έγγραφά μα, λέμε ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και της ε, ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και την ε, ανατολική εταιρική σχέση. Η ερώτησή μου σχετίζεται με έναν ε, πολύ ε, συγκεκριμένο τομέα. Ε, το Erasmus Mundus αποτελεί τρόπο να ενθαρρύνουμε την συνεργασία μεταξύ φοιτητών. Οι φοιτητές έτσι σπουδάζουν μαζί στην Ευρώπη και μεταφέρουν τις αξίες που έχουν μάθει στις πατρίδες τους. Υπάρχει κάποιος τρόπος να αξιολογήσουμε τα ωφέλη αυτού του τύπου της ήπιας συνεργασίας του Εράσμους Μούντους δηλαδή και άλλων τρόπων συνεργασίας ε, φοιτητών και εφόσον προετοιμάζεστε για το 2014-2020 ε, μπορείτε να μας πείτε πώς οι φοιτητέ από την εταιρική, ανατολική εταιρική σχέση θα σπουδάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσοι οι, και πώς φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, σπουδάσουν σε αυτές τις ε, χώρες. Ε, πόσες ομάδες νέων, πόσες μη κυβερνητικές οργανώσεις θα συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Είμαι βέβαιος ότι έχετε τα στοιχεία αυτά. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε μια φωτογραφία της παρούσας κατάστασης και να μας πείτε ποια είναι τα σχέδια σας ε, για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και αναφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτήν την ήπια συνεργασία. Φοιτητικέ ε, ομάδες, οργανώσεις ε, μη κυβερνητικέ κλπ. Ε, οργανώσεις δηλαδή που ε, στηρίζουν ε, τους ανθρώπους στις δραστηριότητες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καθότι οι περισσότερες από τις ερωτήσεις απευθύνονται προς την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα τους δώσω το λόγο. Οι ερωτήσεις αφορούν δύο τομείς. Πρώτον, την, τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής από την, από την εταιρική σχέση και δεύτερον, ε, πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε στο μέλλον και ιδιαίτερα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ακούσουμε ε, τα νούμερα που αφορούν ε, τις πιστώσεις πληρωμών και τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια. Έχω σημειώσει πολλά, θα επικεντρωθώ όμως σε κάποια από τα βασικά θέματα. Καταρχήν, αναφερθώ στις γενικές παρατηρήσεις του κυρίου Γερσπόσκη. Ε, ναι, πράγματι, το θέμα της γενικής ορμής, αλλά και του τελικού στόχου της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας ξεπερνάει τη δική μας εντολή. Ο Επίτροπος Φίλε με τον οποίο συνεργάζομαι ε, σίγουρα θέλει μια όσο γίνεται φιλόδοξη ε, ατζέντα ε, και όσον αφορά τις διατυπώσεις, τη γλώσσα δηλαδή μέχρι τη συνάντηση στο Βίλνιους, ε, αλλά και όσον αφορά τις προτάσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό. Συμπεριλαμβανομένης μια σημαντικής αύξησης στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Επίσης, αν κοιτάξουμε τα στοιχεία του παρόντος δημοσιονομικού πλαισίου, βλέπουμε ότι είμαστε ε, ε, ότι μπορούμε να συγκριθούμε περισσότερο με ε, άλλες αναπτυγμένες χώρες και όχι με προενταξιακές χώρες. 5 τα 100 5 ευρώ κατά κεφαλή, δηλαδή είναι περίπου στις προενταξιακές χώρες δίνουμε μάλλον 50 ευρώ ανά άτομο. Και ακριβώς για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να γίνει ε, μια άμεση σύγκριση ανάμεσα ε, στο πρόγραμμα ΦΑΡ και την ε, παρούσα πολιτική γειτονία. Και ε, ακριβώς επειδή δεν μιλάμε για προενταξιακές χώρες, έχουμε προσπαθήσει να μεγιστοποιήσουμε τη χρηματοδότηση. ώστε να στηρίξουμε τους ε, ανατολικούς μας εταίρους πέρα από τα πλαίσια της ε, ανατολικής ευρωπαϊκής ε, εταιρικής σχέσης. Ε, ναι, ε, κινούμαστε κυρίως με βάση την ε, ζήτηση και ίσως θα πρέπει να αφήσω το θέμα αυτό στους άλλους ομιλητές. Δεν έχουμε πια τεχνική βοήθεια, τεχνική υποστήριξη αυτή καθ' αυτή. Αυτό μάλλον συμπεριλαμβανόταν στην προενταξιακή πολιτική και τότε είχαμε δημιουργήσει μια σειρά από τα μέσα αυτά στα οποία αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες. Ε, αποτελούν αυτά λοιπόν ε, κληρονομιά από τα παρελθόν σε μεγάλο βαθμό ε, και έχουν ενσωματωθεί διάφορες αυτές πτυχέ ε, στα, στους διάφορους φορείς ε, που ε, στόχο έχουν να προωθήσουν τα πράγματα αυτά με βάση τη ζήτηση κυρίω. Ζητώ συγγνώμη διότι νόμιζα ότι είναι προφανές και γνωστό και δεν ήθελα απλά να σας δώσω νούμερα όπως ε, σας είπα, όχι μόνο έχουμε ε, το 100% των ε, πιστώσεων υποχρεώσεων που έχουμε διαθέσει, έχουμε και το 99% των πληρωμών. Και πολύ ευχαριστώ, θα σας υποβάλω τα νούμερα. Αλλά πώς λειτουργεί αυτό. Αν κοιτάξουμε την ε, ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία, είχαμε 2,4 δισεκατομμύρια για την ε, Ανατολή και τον Νότο ε, σε πιστώσεις πληρωμών και είχαμε 1,5 δις για τις πιστώσεις πληρωμών. Θα πρέπει να κοιτάξω αναλυτικά τα στοιχεία, αλλά έχουμε νούμερα μέχρι και το 2012. 700 εκατομμύρια πιστώσεις για την Ανατολή και ένα δις ε, πληρωμές. Η διαφορά ανάμεσα στις πιστώσεις πληρωμών και στις πιστώσεις υποχρεώσεων δεν είναι μόνο η διαφορά στο δυναμικό απορρόφησης, έχει να κάνει και με την ε, εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως ε, γνωρίζει η Επιτροπή σας. Οι πιστώσεις πληρωμών αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστή διαπραγματεύση ε, και είναι πολύ χαμηλότερες από τις ε, πιστώσει ε, υποχρεώσεων. Η διαφορά επίσης εξηγείται από το γεγονός ότι στην αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας είχαμε για το 2011 και 2012 διαφορετικά στοιχεία, οπότε το 2,4 δις ε, δεν έχει ε, ε, μεταφραστεί ακόμα σε πιστώσεις πληρωμών. Όσον αφορά τους μη κρατικού παράγοντες, το, την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια των πυρηνικών και την διαμεθοριακή συνεργασία. Υπάρχουν λοιπόν τα στοιχεία για τους τομείς αυτούς βλέπουμε ότι υπάρχει μέγιστη χρήση ε, των πόρων και η διαφορά ανάμεσα στις ε, υποχρεώσεις και τις πληρωμές αποτελεί συνδυασμό αφενός ε, της μικρότερης διάθεσης για τις πιστώσεις πληρωμών αλλά ε, και λόγω τη ε, συσσόρευση των ε, πρόσθετων προγραμμάτων που εγκρίθηκαν το 2011 και το 2012 που δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί, να το πούμε έτσι, σε πιστώσεις πληρωμών. Μπαίνω στο πειρασμό. Θα μπορούσα να κλείσω βέβαια εδώ πέρα και να ακούσουμε τους άλλους συναδέλφους, αλλά μπαίνω στο πειρασμό να απαντήσω σχετικά με την αρχή more for more και less for less. Μέχρι τώρα προσέξαμε ε, να αποφύγουμε να πούμε ότι το more for more μπορεί να, γίνει, να, το πετύχουμε μόνο ε, τιμωρώντας άλλους. Ε, μπορεί τελικά όσον αφορά το προϋπολογισμό τελικά να είναι ουδέτερη η πρόταση, αλλά εάν δούμε τη νέα πρόταση και την αύξηση του, ε, της χρηματοδότησης, βλέπουμε ότι γίνεται με την πίστη ότι θα πρέπει να υπάρχει θετικό κίνητρο το οποίο να μην ε, προέρχεται μόνο από την μεγαλύτερη αυστηρότητα στα προγράμματα αυτά. Τελικά θα έχουμε συνδυασμό και των δύο. Και τελικά πρόθεσή μας είναι να αυξήσουμε την ε, πρόσθετη χρηματοδότηση που ε, διατίθεται για το More for More στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από τον τελικό προϋπολογισμό που θα διατεθεί ε, και την τελική διατύπωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας όπου οι παράγραφοι για το More for More είναι αυτές που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί στον τριμερή διάλογο. και οι δυο σας αναφέρατε, αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για την ε, Δημοκρατία. Ε, αυτό συνδέεται και με τις εμπειρίες ε, του Ιδρύματος Κονοτάντε Ναόρ στη Λευκορωσία και στις δικές μας εμπειρίες. Ε, πιστεύω ότι το μέσο αυτό καλύπτει ένα κενό το οποίο δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τα παρόντα μέσα με ικανοποιητικό τρόπο δηλαδή να τα χρηματοδοτήσει χωρί να υπονομεύσει την ανάγκη λογοδοσία από τη δική μα πλευρά απέναντι στην ε, αρχή του προπολογισμού. Ε, δηλαδή να μπορέσει να έρθει σε επαφή με μη καταχωρημένες μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, και νέα πολιτικά κόμματα. Κανένα από τα άλλα μέσα δεν θα ήταν αρκετά ευέλικτο μέσο για να το κάνει αυτό. 6 ε, εκατομμύρια έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 3 ε, εκατομμύρια για την Ανατολή και 3 εκατομμύρια για τον Νότο και επιτρέπουμε έτσι στο μέσο αυτό με τη συμμετοχή ε, βουλευτών να μπορεί να αποφασίσει ποια, ε, ποιες ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, και ποια νέα κόμματα θέλει να στηρίξει. Να αναφερθώ λοιπόν και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είμαι πολύ ευγνώμων για την ανάλυση της, του Ιδρύματος Conrad Adenauer. Και θα ήθελα να συνδέσω το θέμα αυτό με το, το θεματολόγιο περί απλοποίησης. Η υποστήριξη της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου για τον δημοσιονομικό ε, κανονισμό που ε, θα τεθεί σε ισχύ από το 2013 θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα θέματα που αναφέρθηκαν. Δηλαδή να έχουμε πολύ περισσότερη ε, υποχρηματοδότηση, μία μη κυβερνητική οργανώση δηλαδή να καλύπτει και άλλες τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις με τις οποίες είναι εύκολο να έχουμε άμεσες επαφές. Και επίσης ε, να επιτρέψει αύξηση του του ορίου. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι μπορούμε να υποβάλουμε το θέμα αυτό στην αρχή του προπολογισμού και ε, με ικανοποίηση σημειώνω ότι μπορέσαμε τουλάχιστον ε, να εξαλείψουμε κάποια από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταίροι μας και επίσης βλέπουμε ότι είναι σημαντικό να συλλέγουμε πάλι τις εμπειρίες μας, να επικαιροποιούμε τα στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα θέματα αυτά ένα θέμα που έχει να κάνει και με αυτό που είπατε εσείς. σημαντικό είναι να μην ε, καταλήξουμε σε, σε μια κατάσταση όπου να δεσπόζουν τα, ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, δεν θέλουμε δηλαδή ε, να φροντίσουμε να μην καταλήξουμε να συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με ευρωπαϊκές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ίσως ε, στην ε, σύμβαση να ήμασταν υπερβολικοί. Θέλαμε ε, οποιαδήποτε οργάνωση χρηματοδοτούμε να έχει στενές σχέσεις με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στις χώρες αυτές. Θα συνεχίσουμε βέβαια να ακολουθούμε τον τρόπο αυτό, αλλά θα φροντίσουμε να μην καταλήξει αυτό να αποτελέσει γραφειοκρατικό άχθος, διοικητικό άχθος. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει από το 2013 και μετά. Η Λευκορωσία είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες ε, για να βρούμε τη σωστή ισορροπία ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις επαφές μας με την ε, παρούσα κυβέρνηση, μεγιστοποιώντας ε, την υποστήριξή μας προς τις τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και την διασπορά. Και Ε, αυτό αποτελεί μία από τις ε, απαντήσεις μας όσον αφορά την Ανατολή. Και Επίση, φροντίσαμε να συνεχίσουμε να είμαστε σε πολύ στενή επαφή με του δικαιούχου εδώ στι Βρυξέλλε. Κάθε έξι μήνε, λοιπόν, συναντώμαστε με εσά και με πολλού από του εταίρου σα, προσπαθώντα ε, να διαδώσουμε τι βέλτιστε πρακτικέ. Θα κλείσω εδώ, διότι μα πιέζει ο χρόνο. Ο χρόνο μπορεί να υπάρξουν και άλλε παρατηρήσει και ερωτήσει ε, ευχαριστώ όμω θα σας απαντήσω και σε όλα τα άλλα πράγματα που σημείωσα. Ευχαριστώ. Ρίτσαρτ, θέλεις να προσθέσεις κάτι. Ε, ε Τέθηκε μια σε σχέση με, με το έρασμα και τη στήριξη για τους ε, φοιτητές. Μπορείς, Ρίτσαρντ, λοιπόν, να απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήματα έμειναν αναπάντητα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να πω ότι η ερώτηση για η αμφισβήτηση μάλλον του πόσο πολιτικά οθούμενη ήταν η στήριξη προς την ανατολική εταιρική σχέση, εγώ πρέπει να πω ότι αμφισβητώ. Είναι από τις ε, περιοχές όπου μας ενδιαφέρει περισσότερο η πολιτική ε, κατάσταση. Έχουμε τις νέες συμφωνίες που ε, θέλουμε να συνάψουμε και θα είναι ατζέντες για την σύνδεση και Ούτως ή άλλως πρόκειται για χώρες που θέλουμε να αναλάβουν και να δεσμευθούν με τις προτεραιότητες κλειδιά σε αυτές τις τη διατάξεις της σύνδεσης. Πιστεύω δηλαδή πως η δική μας προσέγγιση καθοδηγείται από την πολιτική και κάτι που ξέχασα να αναφέρω στις μου, στην αρχική μου δήλωση ήταν ε, ότι η σταδιακή αποχώρηση από τη διμερή βοήθεια της Ρωσίας θα πρέπει να διευκολύνει την ορατότητα για τη δική μας χρηματοδότηση γιατί το μέσο γετνίασης θα εστιάσει περισσότερο το ανατολικό τμήμα του θα εστιάσει περισσότερο στις εταιρικές σχέσεις και έτσι θα διευκολυνθεί πιστεύω το θέμα που αφορά τα νούμερα και πώς μπορούμε να καταστήσουμε σαφές στις χώρες εταίρους μας τη στήριξη που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα μόρφο μόρο, ο Μάρκος είπε κάποια παραπάνω πράγματα. Υπάρχουν τρόποι με τον οποίο μπορείς να προβλέψεις ευελιξία μέσα από, κατά τη διάρκεια μάλλον της προγραμματικής περίοδου που μπορεί να επιτρέψει και βελτιώσεις, αλλαγές με βάση την απόδοση. Ορισμένοι μπορεί να θεωρούν πως κέρδισαν ενώ άλλοι πως έχασαν, αλλά... Εάν χρησιμοποιήσουμε την, ε, τα μέσα ευελιξίας όπως το φουχσέτ στις ε, κατανομές, θα μπορούσαμε όντως να ε, το ελέγξουμε. Κάτι επίσης που δεν ανέφερα στην αρχική μου εισήγηση ήταν η σημασία της, για την ανατολική εταιρική σχέση η σημασία της συμβολής που θα γίνει στο πρόγραμμα ράσμους για όλους στο μέλλον. Θα είναι ένα ένας εξαιρετικά σημαντικός μηχανισμός για να μπορέσουμε να φτάσουμε ευρύτερα στην κοινωνία και κυρίως στη νέα γενιά. Δεν μπορώ βεβαίως να σας δώσω νούμερα για τον αριθμό των φοιτητών που θα ωφεληθούν στο μέλλον. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του κονδυλίου που θα δοθεί Στον οδικό χάρτη για την Ανατολική Εταιρική Σχέση είχαμε έναν αριθμό στόχο για τον αριθμό δηλαδή των φοιτητών που θα ωφεληθούν από το Erasmus Mundus το 2012 και 2013 και μπορώ να σας στείλω κύριε Ευρωβουλευτά το νούμερο μετά. Θα πρέπει να σας πω πως ε, σήμερα το πρωί σας ε, έκανα μια προειδοποίηση όσον αφορά τον βαθύτερη σχεδιασμό για το μέλλον και τον προγραμματισμό και το ήδη είπα όταν δέχτηκα να έρθω σήμερα καθώς πρόκειται για μια λεπτή διαδικασία που οδηγεί προς την περίοδο 2014 με 20 να είστε βέβαιοι πως πολλή εσωτερική εργασία γίνεται και έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά έχει γίνει για το διμερές πρόγραμμα με τις ε, αντιπροσωπείες της Ένωσης Επιτόπου, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εντοπισμό των τομέων κλειδιών που θέλουμε να ε, δουλέψουμε με τους εταίρους μας τη νέα δημοσιονομική περίοδο. Αλλά δεδομένου ότι επικρατεί αβεβαιότητα για τον προϋπολογισμό και για το πώς θα οριστικοποιηθούν οι ρυθμίσεις more for more τις επόμενες εβδομάδες είναι δύσκολο να μπούμε σε περιβολικά πολλές λεπτομέρειες για τους προγραμματικούς μας στόχους σήμερα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτές τις απαντήσεις. Σιδωνία, μάλλον θα πρέπει τώρα να συνοψίσεις για να κλείσουμε και τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω την συζήτηση, εκτός και αν κάποιος άλλος από τους προσκεκλημένους μας θέλει να ε, προσθέσει κάτι. Όχι, νομίζω πως οι περισσότερες ερωτήσεις απευθύνονταν στα δύο θεσμικά όργανα. Ωραία, λοιπόν, τότε να προχωρήσω προς την ε, ε, σύνοψη. Είμαι ευτυχής που έγινε αυτή η σημερινή συνεδρίαση, αν και πολλά από τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, γιατί ξεκίνησε μια διαδικασία ε, ανταλλαγής απόψεων, θα τη συνεχίσουμε. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω έναν γενικότερο λόγο για τον οποίο γίνεται τέτοια συνεδρίαση όπως σήμερα και γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν θέλουμε να ικανοποιήσουμε απλά την περιέργεια κάποιων. Δεν θέλουμε απλά να ανακυκλώσουμε διαθέσιμα ή μη ε, δεδομένα. Πρόκειται για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα χρήματα των φορολογουμένων. Κάποιες φορές ε, είμαστε επιπισμένοι πως τα όσα κάνουμε ε, είναι σωστά, αλλά δεν είναι αυτό απαραίτητα σαφές για τον ναι, απλό κόσμο. Και είναι καθήκον μας και ευθύνη μας να αξιολογήσουμε τι κάνει η Ένωση όσον αφορά την επίτευξη πολιτικών στόχων, αλλά και όσον αφορά την λογοδοσία και τη διαφάνεια. Θα με λοιπόν να είμαστε μόνο αμυντικοί για να μας πούν όλοι δηλαδή όλα όσα κάνουμε είναι καλά για, απλά και μόνο επειδή εμείς τα κάνουμε πρέπει να μπούμε σε βάθος γιατί υπάρχουν ε, όλα ένα και περισσότερες ανησυχίες όσον αφορά την ανάπτυξη της δημοκρατίας και τον τρόπο με τον οποίο οι έξι χώρες της ανατολικής ε, αυτής συνεργασίας ε, διοικούνται. Και αυτό θα αφισβητήσει και τα ευρωπαϊκά χρήματα. Τα, όλο ένα και περισσότερο θα πρέπει να δούμε τι, τι γίνεται με εκείνα τα χρήματα που πάνε άμεσα στον εθνικό προπολογισμό αυτών των κρατών, εφόσον υπάρχουν ανησυχίε για τη δημοκρατία και το επίπεδο τη διαφθορά. Πιστεύω λοιπόν πω από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να παρακολουθούμε τι εξελίξει ώστε να εξασφαλίσουμε σε κάθε στάδιο, στο επίπεδο νομοθεσίας, στο επίπεδο εφαρμογής, πως τελικά τα χρήματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αξίες της Ένωσης και όχι αντίθετα προς αυτές. Δεν ε, είναι μόνο λοιπόν τα νούμερα και οι σωστοί λογαριασμοί, αλλά ε, θέλουμε να έχουμε αυτά τα λιγοστά χρήματα, που είναι τελικά λιγοστά, να είναι σωστά στοχοθετημένα. Και πρέπει να συνεργαστούμε ως ευρωβουλευτές, αλλά και ως εκτελεστικό της Ένωσης και στόχο να έχουμε να μπορούμε να λογοδοτήσουμε για αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και επιμένω και πάλι για να μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία όσο μπορεί περισσότερο για να μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε σε αυτό το καθήκον ελέγχου που έχουμε, Για διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο να δίνουμε τη συγκατάθεσή μας και να έχουμε την πολιτική βούληση να συνεχίζουμε και να το καθιστούμε κατανοητό στους πολίτες. Για ποιο λόγο δηλαδή ασχολείται οικονομικά, εμπλέκεται οικονομικά η Ένωση στις χώρες της Ανατολικής ε, γειτονίας. Σήμερα μιλάμε για την Ανατολική εταιρική σχέση, αλλά το ίδιο πράγμα ισχύει και για τη Νότια ε, γειτονιά ε, πρέπει σε κάθε φάση να υπάρχει έλεγχος και να εξασφαλίζεται διαφάνεια και η πλήρης λογοδοσία για τα όσα κάνουμε ως Ένωση. Και τώρα θα συνεχίσω λοιπόν τις ε, ανταλλαγές ε, απόψεων και στοιχείων με την Κομισιόν ώστε να διευκρινιστούν όλα αυτά τα στοιχεία και θα τα συμπεριλάβω σε αυτή τη δημοσίευση που θέλουμε να κάνουμε Επειδή ο συνάδελφος ανέφερε το έρασμος για όλους και το ανέφερε και ο κύριος Τίμπελς, εμένα ανησυχούν κάποιες εξελίξεις σε αυτόν τον κανονισμό, που είναι μια καλή, ε, ένα καλό παράδειγμα για να το μελετήσουμε. Ξέρω πώς είναι στον τριμερή διάλογο, ξέρω πώς είναι η υποδιαπραγμάτευση, αλλά από την άποψη του προπολογισμού βλέπω κάποια προβλήματα για την εφαρμογή σπουδαίων πολιτικών ιδεών. Και πιο συγκεκριμένα, έρασμος για όλους. Η ιδέα είναι να υπάρχουν τα χρήματα και το πρόγραμμα και να εφαρμόζονται τα προγράμματα αυτά από τι χώρε τι γειτονικέ. Εγώ φοβάμαι πω οι φοιτητέ θα υποφέρουν. Έχω πολύ σοβαρέ αμφιβολίες για, το, για τις ικανο, ικανότητες των χωρών αυτών να τα επεξεργαστούν όλα αυτά δηλαδή, να εξυπηρετηθούν σωστά οι φοιτητέ, γιατί είναι οι υπηρεσίε τη Κομισιόν που τα διαχειρίζει. Δεν ξέρω ακριβώ ποιο κάνει, πάντω γίνεται πιο κεντρικά. Και η αποκέντρωση, μόνο και μόνο προς χάρη της αποκέντρωση δεν ε, ε, είναι σίγουρο πως θα βγει σε καλό. Γιατί ξέρω πως ε, και για χώρες που έχουν πολλά παρεδώσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παιδεία και τον πολιτισμό έχουν επενδύσει πολλά Και σίγουρα δεν είναι εύκολη η διαδικασία για να δοθούν τα χρήματα στα πανεπιστήμια και στους φοιτητές. Το να τα δώσουμε λοιπόν τα χρήματα χωρίς να τους προετοιμάσουμε τις χώρες εταίρους ε, μπορεί τελικά να δυσχεράνει την κατάσταση για τους φοιτητές και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε πως ε, οι υποτροφίε αυτέ θα πρέπει να δίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πραγματικά. Γιατί ούτω ή άλλως όλα αυτά τα χρήματα που στόχο έχουν τις χώρες της Ανατολικής Γετνίασης θα πρέπει να ωφελούν τον κόσμο που ζει εκεί. Όχι απλά και μόνο να είμαστε εμεί ήσυχοι ότι κάνουμε τη δουλειά μα καλά. Δεν αρκεί αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να χρησιμοποιούνται τα χρήματα από όσο γίνεται περισσότερους και να ωφελήσουν τον κόσμο που ζει εκεί. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με αυτή τη συνεχιζόμενη προσπάθεια και ευχαριστώ τους ε, προσκεκλημένους μας που ήταν ε, ε, έτοιμοι να έρθουν εδώ να μας ακούσουν και να μας ενημερώσουν και να συνεχίσουμε το διάλογο. Ευχαριστώ Σιδωνία. Να προσθέσω μόνο ότι συμφωνώ με την Σιδωνία ότι δηλαδή Όντω πρόκειται για την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου για το πώς και πού δαπανώνται τα χρήματά μας. Και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Να ζητήσω συγγνώμη στου προσκεκλημένους ότι, ε, που θεώρησαν ότι μπορεί να μπορούσαν να θέσουν ερωτήσεις, αλλά αυτή είναι μια συνεδρίαση του προπολογισμού και οι ευρωβουλευτές πρέπει να είναι σε θέση να θέσουν ερωτήσεις. Ε, Ζητώ συγγνώμη αν παραπλανηθήκατε, αλλά έτσι έχουν οι κανόνες. Δεν είναι ανοιχτή η ακρόαση, είναι συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών. Αυτά λοιπόν για την πρωινή μας συνεδρίαση. Κλείνουμε εδώ και ελπίζω να σας ξαναδώ όλους τις τρεις και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που συνέβαλαν στην εξαίρετη αυτή συνεδρίαση.